είχαμε... Χάσατε δύο πλοία μετά από δύσκολες συνθήκες. Ελπίζουμε η Κομισιόν να ε, μπορέσει να αναλάβει μια δράση και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Τεχέιρα. Φρανσίσκο Τεχέιρα λέγουμε. Η οργάνωση παραγωγών που εκπροσωπώ λέγεται το Οργάνωση Παραγών του λιμένου και του ποταμόκολπου του Μαρίνη, το πρωμάδα Αναγνωρίστηκε ως αντιπροσωπευτική οργάνωση το 1986 με εδαφική αρμοδιότητα την περιοχή της Ποντεβέδα για τις δραστηριότητε, στην περιοχή του, στην παράκτη περιοχή τη Ισπανία και τη Πορτογαλία που ασκούν δραστηριότητε νοπών προϊόντων. Επίση χρησιμοποιούν και άλλα λιμάνια τη περιοχή τη Γαλλικία για τη δραστηριότητα του. Η οργάνωση είναι μία από τι 7 οργανώσει παραγωγών που αναγνωρίζονται από την αυτόνομη περιφέρεια της Γαλλικίας και τα, η παραγωγή των, των οποίων ασκούν δραστηριότητα νοπών προϊόντων. Ένας κοινό παράγοντα για όλες αυτέ τι οργανώσεις παραγωγών είναι ο τύπος σκάφους με έναν αριθμό ναυτικών από 9 έως 12 που ανήκουν σε μια επιχείρηση μικρών διαστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό της ΕΛΙΕΣ ε, δεν απαιτείται να υπάρχει μια υψηλή χρηματοδότηση επιχειρήσης για μεγάλες επενδύσεις, αλλά ε, σημαντική είναι η συνεισφορά της γνώσης και η γνώση του επαγγέλματος ναυτικού. Ε, οι, τα ποιοί ναυτικοί που προσπαθούν να βελτιώνουν και να επενδύουν στην θάλασσα με μικρά εισοδήματα. Είναι ένας ε, κλάδος πολύ επαγγελματοποιημένος, ε, δραστηριοποιείται με παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνει αποτελεσματικές, ε, έχει αποτελεσματική απόδοση προσφέροντας ε, καλά σκάφη, καλούς ναυτικούς και που βασίζεται σε μια συμμετοχή των ναυτικών στο ποσοστό των πωλήσεων των ε, αλλιευμάτων Ολοκληρώνοντα έτσι την ευθύνη μέσα στον κύκλο της επαγγελματική δραστηριότητα, Η βιωσιμότητα και η συνέχεια κάθε της όπω όπως και των ελεκτικών επιχειρήσεων, βασίζεται σε μια οικονομική αποδοτικότητα αν βγάλουμε τις δαπάνες, ε, μάλλον ε, με την, ε, πρέπει μετά την εξισορρόψη εσόδων-εξόδων υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να υπάρξουν νέες επενδύσεις. Οι δαπάνες δραστηριότητε των επιχειρήσεων αυτών είναι αυτές που χρειάζονται για την παραγωγή και θέση πρώτη πώληση. Μεταξύ αυτών είναι οι μισθολογικές δαπάνες, οι σφορές, per ε, ε, η, αγορά προϊόντων ε, του υλικού της ελίας, δίκτυα, καλώδια και λοιπά, η προετοιμασία και η συντήρηση, η, αποβίβαση και η, η εκφωτωση η συσκευασία. Στο τελευταίο τμήμα των δαπανών που είναι τα καύσιμα είχαμε μια δύσκολη αρνητική εξέλιξη από την ε, από τα τελευταία χρόνια λόγω των, υψη, των μεγάλων αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, ιδίως μετά το 2004, που είχαν ανετικέ συνέπειες στην οικονομική ισορροπία των λογαριασμών μας. Τα έσοδα προκύρχονται από την πρώτη πώληση των, ε, από, των ε, προϊόντων στις αγορές, στις αλευτικές αγορές, στα εγκεκριμένα κέντρα, μέσω ενός συστήματος ε, μειοδοτικών διαγωνισμών. Στις, ε, στις αγορές συγκεντρώνονται τα προϊόντα από διάφορα πλοία που βασίζονται σε, ε, στηρίζονται στην ανάγκη να υπάρχουν τιμές σε, καλές, ε, σε καλές τιμές των προϊόντων. Τα παραδοσιακά συστήματα πώληση των ψαριών μέσω των μειοδοτικών διαγωνισμών δεν επιτρέπουν στους παραγωγούς να περάσουν το κόστος εκμετάλλευσης παραγωγής ε, ε όπως έπρεπε. Οι δαπάνες πρώτης πώληση παρέμειναν σε σταθερές τιμές, μεταξύ των οποίων και σε στιγμές κατά τις οποίες καταγράφηκαν ε, διαφο, διαφοροποιημένες, διαφοροποιήσεις των τιμών ε, του, των καυσίμων. Κάτι που επέτρεψε ε, οι χαμηλές τιμές παροτρύνει τώρα τους ε, ψαράδες να παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες, κάτι που ε, οδηγεί ωστόσο σε μείωση της απόδοσης και αυξάνει το, τα κίνητρα για υπεραλίευση. Ωστόσο, ο κλάδο εκτιμά μια, ολοένα και μεγαλύτερη, ένα ολοένα και μεγαλύτερο περιθώριο για την δημιουργία τη αλυσίδα αξία των προϊόντων τη αλία από το ξεκίνημα μέχρι το τελικό καταναλωτή χωρί να μπορεί να μεταποιηθεί το αλληλευτικό προϊόν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η διανομή των αλληλευμάτων της ε, του κοινοτικού στόλου ε, νοπών προϊόντων μέχρι να φτάσει στον καταναλωτό πήγαινε στην, βασιζόταν σε ανταγωνιστικό μεταξύ των ε, διαφόρων αγορών. Τι αγορέ προέλευση, τα μικρά λιμάνια όπου γίνονται οι αποβάσει των αλλιευμάτων και η πρώτη πώλησή του, τα, η αγορά σε χονδρική όπου βρίσκονται οι επιχειρηματίε του κλάδου και συναντιούνται με, με τις αρχικές αγορές καθώς και τις μεταποιήσεις για να μπορέσουν να διανύμουν κατόπιν στο λιανεμπόριο και την τρίτη αγορά, την αγορά την, της, το λιανεμπόριο στο οποίο ε, ο καταναλωτής φτάνει στην αγορά του προϊόντος. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 η αγορά άλλαξε σημαντικά και άλλαξε ολόκληρος ο πρωτογενής κοινοτικός παραγωγός αλίας ε, για πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στους εξής. Βελτίωση επιμελητιακού χαρακτήρα, δηλαδή εξελίσσονται οι υποδομές μεταφορών είτε οδικέ είτε θαλάσσιες ή κυριω ε, εναερίε. Ε, οπότε το προϊόν μπορεί να έρθει από πολλές περιοχές του κόσμου σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάτω από καλε τεχνικές συνθήκες. Επίσης άλλαξαν οι συνηθειε του καναλωτή, μορφή, τοπο περιοδικότητα αγοράς, χρόνος για την αγορά, απέτηση νέων μορφών παρουσίας και καταναλωτή των προϊόντων, αλλά και ενσωμάτωση και ε, σούπερ μάρκετ ε, και μεγάλων αλυσίδων τροφίμων. Αυτές οι αλλαγές δημιούργησαν νέα κύκλους διανομής και τροφοδοσίας, δημιουργώντας ένα παράλληλο ε, διάβλο από τον παραδοσιακό. Επίσης γίνονται απευθείας πωλήσει στο κοινό και μπορούν να προκληθούν αλλαγές στη ζήτηση και στη συνήθεια του καταναλωτή. Η άμεση εισαγωγή δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις κεντρικές αγορές, επηρεάζοντας με τη σειρά και τις ε, ε, αρχικές αγορές. Όταν γίνεται η αγορά στα λιμάνια, δημιουργήθηκε και, μια μεγαλύτερη, και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός στις αγορές προέλευσης. Και επιπλέον υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική και διαχειριστική ικανότητα που επιτρέπει μείωση του κόστους και μεγαλύτερα περιθώρια. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο ταυτόχρονα, παρενθετικά τα τρόφιμα, μάλλον στο, στα τρόφιμα, το φθηνό δεν είναι πάντα το, το καλύτερο. Ίσως η, η υψηλή δυνατότητα αγοράς της κοινωτικής αγοράς επιτρέπει να αγοράζονται προϊόντα ε, από τρίτες χώρες ε, σε χαμηλότερη τιμή, ωστόσο οι εργαζόμενοι ε, στον τομέα της ε, στον τομέα αυτό δεν μπορούν να ανταγωνιστούν γιατί μερικές φορές η μεταφορά είναι ακριβότερη από το προϊόν. Με αυτή τη μικρή, μετά από αυτή τη μικρή ανάλυση της κατάστασης του κλάδου στο, στην παραγωγή αλίας ενώπων προϊόντων, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν προλάβαμε, δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές της αγορές. Ωστόσο θα πρέπει όλοι, έπρεπε όλοι να βρούμε μια νέα ισορροπία και να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ασκούμε με αξιοπρέπεια το επάγγελμα, κάνοντας μια βιώσιμη αλληλεία από την οπτική γωνία των βιολογικών πόρων και της οικονομικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο, ενός, ε, στο πλαίσιο διαφάνειας, ασφάλειας τροφίμων και των καταναλωτών, δίνοντας μία δίνοντας δυνατότητα να κερδίζουν ε, τα επαρκή σε αυτή τη δύσκολη και πολύ απαιτητική δουλειά. Η κατάσταση του κοινοτικού στόλου σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες, ε, που έχουμε, τις επιτυχίες μας στην ασφάλεια της θάλασσας, τις ευτυχές εργασίες, δικαιώματα των εργαζομένων, ποιότητα των προϊόντων κτλ. δεν θα πρέπει να χαθούν από την οπτική μας. Και είναι υποχρέωση όλων να δώσουμε μια συνέχεια στις πολιτικές αυτές. Υπάρχει περιθώριο μεταξύ των τιμών της πρώτης πώληση και των τιμών για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχεια χωρίς να υπάρξει καμία μείωση των εγγυήσεων προς τον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα της αλληλείας και τη βελτίωση των ε, αποθεμάτων και των πόρων. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους συνέχεια έναν ε, στον κλάδο, στα πλαίσια μιας κοινή οργάνωσης αγοράς, νομίζω ότι ο οργανώσεις παραγωγών είναι ο μόνος διαμεσολαβητής που θα μπορούσε να ε, συγκεντρώσει τους παραγωγούς και να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή προσθέμενης αξίας των προϊόντων μας στην αλυσίδα αξίας. Αυτό που λέμε κλείνουμε τον κύκλο της από τη θάλασσα μέχρι το τραπέζι θα πρέπει να είναι πρόκληση και στόχος όλων. Σε αυτή την περίοδο γενικής κρίσης, ωστόσο, είναι δύσκολο να υπάρξουν συλλογικά μέτρα που θα αλλάζουν ριζικά την ε, σημερινή εικόνα του τι κάνουν σήμερα και τι μπορούν να κάνουν οι αλληλείς αλλά είναι αναγκαίο για να προχωρήσουμε και να αναλύσουμε κάποιες δυσκολίες ή αδυναμίες που εμπεριέχουν οι στόχοι αυτοί και μεταξύ αυτών θα μπορούσα να αναφέρω την εξατομίκευση των αλλιευτικών επιχειρήσεων. Πολλά σκάφη με διαφορετικούς τρόπους αλλιείας, παρασυρώμενα πλάδια, παραγάδι κλπ. που λειτουργούν σε διάφορα λιμάνια και διαχειρίζονται πολλές ε, επιχειρήσεις, κάνουν δύσκολο να υιοθετηθούν σε κοινά μέτρα. Υπάρχουν μικροί οικονομικοί πόροι. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και των οργανώσεων παραγωγών δυσχεραίνουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του απαραίτητου κεφαλαίου για να προσαρμοστούν στις νέες συμβάσεις που απαιτούν οι διανομή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επίσης μικρή γνώση των μηχανισμών και των αγορών που είναι διαφορετικές από τις αγορές προέλευσης. Υπάρχει πολύ χαμηλή εμπορική εμπειρία για, τη μεταποίηση των προϊόντων. Η κατάσταση των πόρων, ο, ο στόλο σε, ε, ε, αλλιεύει σε κοινοτικά ύδατα και υφίσταται μια σειρά ε, ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Τα κριτήρια ανάθεσης των ποσοστώσεων συγκεκριμένων ε, ειδών ε, την χάνει κοινή διαφήμιση. Δεν υπάρχει ωστόσο ατομική ποσόστοση, άρα αυτό δυσχεραίνει τη διαχείριση των προγραμμάτων αλίας. Όταν ολοκληρώνεται η ποσόστοση, σταματάει η αλία για όλους, ανεξάρτητα αν κάποιο είχε κάνει μεγάλη μικρή αλίευση. Όπως είπαμε νωρίτερα, οι οργανώσει παραγωγών θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν αυτού του στόχου και αυτέ τι προσκλήσει, Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, Ζητούμε να υπάρχουν βελτιώσεις στην νομοθεσία που θα επιτρέπει να αναλυφθούν οι δυσκολίες και να ε, βελτιωθεί η χρηματοδότηση των οργανώσεων και η βελτίωση των μηχανισμών παρέμβασης που έχουν αυτή τη στιγμή όταν ε, με δυνατότητα να πως μειώνονται οι παραγωγοί όταν μειώνεται το, ο, ο, των, του, των ε, ειδών. Οι οργανώσει παραγωγών θα πρέπει να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο για την εξασφάλιση μια ορθολογική διαχείριση τη αλληλεία και βελτίωση των συνδικών πώληση και παραγωγή, εξασφαλίζοντα εισοδήματα στου παραγωγού και εξασφαλίζοντα στου καταναλωτέ και ποιότητα και διαφάνεια για τα πρώτα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ενισχυθούν στο εσωτερικό των κοινών οργανώσεων αγορά οι δομέ αυτέ για να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του και να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση ώστε να βελτιωθούν οι ανθρώπινοι πόροι των οργανώσεων παραγωγών μέσω της περίληψης αυτούς ειδικών στην εμπορία, στην τεχνολογία τροφίμων, βιολόγων, ε, ε, υπευθύνων δημοσίων σχέσεων, να ενισχυθούν η λειτουργία των νέων και των παλιών οργανώσεων για να ε, ενισχυθεί η επιθυμία συμμετοχής και η συμμετοχή στο μεγαλύτερο ε, στόλο συλλογικών έργων και βελτιώνοντας και τα ε, λειτουργικά προγράμματα. Η βελτίωση των σημείων υποδοχής των νέων προϊόντων στις αγορές, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανείχνευσης, ομοιογένεια και επαλήφθηση ποιότητα των προϊόντων. Η βελτίωση των συστημάτων χρηματοδότηση του κεφαλαίου για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι αυξήσει στι δαπάνε προσωπικού και ε, χωρί να επιβαρύνονται οι πελάτε. Μηχανισμοί παρέμβαση. Η τιμή των προϊόντων τη Ελία επηρεάζεται από, την από το υψηλό ποσοστό των εισαγόμενων προϊόντων το σημερινό σύστημα των ε, ε, αντισταθμιστικών πρημοδοτήσεων για την παρέμβαση στα προϊόντα με τιμές ε, μικρότερες από την απόσυρση για, για την ελίευση νοπών προϊόντων αναφέρεται στο παράδειγμα 6 στο παράδειγμα 4 του κανονισμού 104-2000 και συμπεριλαμβάνει μια σειρά από είδη τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επικυροποίησης και να υπάρξουν και να σωματωθούν και νέα προϊόντα τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη τότε. Επίσης, οι διαδικασίες μεταποίησης για τις ενισχύσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 23 του κανονισμού 104-2000 πρέπει και αυτέ να επικαιροποιηθούν και να υπάρξουν νέε λύσει ε, όσον αφορά ορισμένε ποιότητε προϊόντων. Σήμερα μπορούν να γίνουν εισαγωγέ των προϊόντων με την επιλογή εφαρμογή μηχανισμών ε, αντιστάθμιση με τιμέ κάτω από τι τιμέ απόσυρση. Οι εισαγωγέ πραγματοποιούνται, αλλά ε, θα καταργηθεί το το όφελος από το συγκεκριμένο τελωνιακό καθεστώς ε, για τις ενολόγω ε, ποσότητες. Επίσης, οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να καθορίζουν και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα μηχανισμούς περιορισμού των εκφορτώσεων, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερες ε, εισαγωγές. Ε, ε, διότι και με αυτόν τον τρόπο ε, δεν μπορεί να καταστήσει δυνατό ο στόχο μείωση τη προσφορά. Επίση, θα ήθελα συντομία να σα αναφέρω δύο λόγια για το σχέδιο το οποίο αναπτύσσουμε εμεί ως οργάνωση παραγωγών το 2007 και το οποίο στοχεύει ε, βελτίωση της ποιότητα των αλληλευτικών προϊόντων. Με χρηματοδότηση της αυτόνομης περιφέρειας της Γαλλικία στα πλαίσια των ενισχύσεων του, του Ταμείου Ολία, το που θα ολοκληρωθεί το 2010 με την συμμετοχή 12 αλληλευτικών μονάδων συνειδητοποιούμε το μικρό αριθμό των ε, ε, αλλιευμάτων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς επίσης και τη μεγάλη ποικιλομορφία των ειδών. Ε, αλλά δεν μπορούμε να ε, παραμείνουμε αδρανείς, γιατί, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ωφελήσει καθόλου τις προοπτικές μας. Το σχέδιο αποτελείται από την έγκριση μια σειρά τεχνολογικών επενδύσεων ε, στις, σε 12 αλλιευτικές μονάδες, μαζί με εν πλώ, μαζί με επενδύσεις στην ξηρά. σε ένα σημείο ελέγχου και επαλήθευση στην Ιχθυροσκάλα Μαρίν. Εδώ ε, πρέπει να προσθέσουμε διάφορα σεμινάρια κατάρτιση για τι νέε τεχνολογίε ε, του προσωπικού εμπλό, καθώ επίση η διάδοση ε, και η κατανόηση των κοινών κανόνων τυποποίηση των λευτικών προϊόντων, καθώ επίση και τη μορφολογία και του βάρου των δοχείων. Όσον αφορά τι επενδύσει εμπλό, εδώ μιλάμε για την εγκατάσταση ψηφιακή ζυγαριά ε, και εκτυπωτή, έτσι ώστε να έχουμε σήμανση που να πληρεί όλα τα πρότυπα, συμπεριλαμβάνοντα την κωδικοποίηση με γραμμικό κώδικα, ε, καθώ επίση ε, και διάφορου μηχανισμού εντοπισμού που επιτρέπουν την ανάγνωση με τι νέε τεχνολογίε ραδιοσυχνότητα. Φορητό υπολογιστή και υπολογιστή αφή στο χώρο διαλογή αλλιεύματων, όπου θα υπάρχει διαχείριση ενό λογισμικού, λαμβάνοντα υπόψη τα πρότυπα ε, τα πρότυπα τυποποίηση των προϊόντων και το βάρος ε, στις ε, συσκευασίε. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερες πληροφορίες προς τον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα ημερομηνία και ώρα αλλίευση και εδώ λαμβάνεται υπόψη η θέση που δείχνει το GPS. Ζώνη αλλίας αναφέροντας περισσότερα στοιχεία για το πού βρίσκονται οι ζώνες αυτές. Συγγνώμη που σας ε, διακόπτω, πρέπει να τελειώσετε γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, όνομα... τελειώνω, τελειώνω Πρόεδρε. Όνομα ε, σκάφους, ε, ε, στοιχεία που έχουν να κάνουν με, την, με τα στοιχεία που έδωσε η ζυγαριά κτλ. Ε, και εδώ ε, μιλάμε για μια τεχνολογία που είναι πολύ παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται ε, από τα πιο εξελιγμένα σκάφη για να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα και ποιότητα των προϊόντων. Ε, αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μιλήσατε για ορισμένες πτυχές του ε, κανονισμού που θα πρέπει να αλλάξουν και νομίζω ότι αυτά θα μπορούσαν να σημεύσουν για την συζήτηση εν ώψη της μελλοντική μεταρρύθμισης. Για 15 λεπτά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ζακ Πισόν, ο οποίος είναι διευθυντής ε, της ε, ε οργάνωσης αλλιέων ε, στην ε, περιοχή στην περιοχή της Μάνχης. Λοιπόν, λύσαμε τα τεχνικά προβλήματα και πάμε τώρα στον επόμενο μιλητή, στον δόκτωρα Ματία Κελερ. Ε, τον γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Επιτροπή μας, εκπρόσωπος της οργάνωσης των μεταποιητών και των... Α, και, εδώ θέλουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όχι, τι θα κάνουμε τώρα. Ε, η σύγχρονη τεχνολογία τελικά μας καθυστερεί τις εργασίες. Ποιο μπορεί να μιλήσει χωρί υπολογιστή να σηκώσει το χέρι του. Ο κύριο Στίβενσον, τέλεια, βρήκαμε κάποιον ομιλητή. Ο κύριο Στίβενσον, πρόεδρο ε, τη οργάνωση Αλλιών τη Σκωτία. Κύριε Στίβενσον, ε, λυπάμαι που δεν είναι και ο συνάδελφό από τη Σκωτία που θα πρέπει να σήμερα, από έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα Αξιότιμοι βουλευτέ, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ στην Επιτροπή σα. Καταρχά, να συστηθώ. Ονομάζομαι Ρόμπερτ Στίβενσον και είμαι επικεφαλή ε, τη οργάνωση παραγωγών τη ε, Σκοτία, μια ε, οργάνωση παραγωγών αλλιέων, η οποία γνωρίζεται από την Ένωση. Βρισκόμαστε στη Σκοτία, στο Πίτερχετ και βασικά ασχολούμαστε με τα λευκά ψάρια, το γάδο, το εγκλεφίνο και εκπροσωπώ την ε, Σκοτική Ένωση Παραγωγών Εχθείων που περιλαμβάνει και τις 10 οργανώσεις στη Σκοτία. Βασικά ασχολούμαστε με τα αλλιεύματα, την ε, διαχείριση και την εφαρμογή των ε, σχεδίων ελάχιστης τιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο και την διαχείριση των ποσοστώσεων που δίνεται από την κυβέρνησή μας. Το 1999 οι σκοτικές ε, οργανώσεις ε, δημιούργησαν την οργάνωση Seafood Scotland, η οποία αναλαμβάνει τις εξωτερικές ε, λειτουργίες και ενέργειες marketing εξ ονόματος των οργανώσεων παραγωγών ηχθείων στη Σκωτία. Και μία από τις πρώτες τέτοιες πρωτοβουλίες μας ήταν να αναπτύξουμε ένα σχέδιο υπεύθυνης αλληλείας για την τήρηση βασικών ε, προτύπων υγιεινής. Και υπάρχει αναφορά επίσης στα στάνταρ, στα πρότυπα MSC, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τρέχον έτος. Αφιερώσαμε σημαντικούς πόρους ε, στην ε, συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων για να διατηρηθούν τα επίπεδα τιμών σε ό,τι αφορά και τα τρέχοντα έξοδα για τη συντήρηση των σκαφών, σε ό,τι αφορά και τα έξοδα καυσίμων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά φθηνά υποκατάστατα ψαριών, όπως τα ονομάζουμε, όπως ο Παγκάσιος και το Τιλάπια. Φυσικά, περιορίζω, είμαστε υποχρεωμένοι να μην πουλάμε κάτω από τις ελάχιστες τιμές. Ωστόσο, πολλές από τις ελάχιστες τιμές αυτές δεν ισχύουν σε κάποια είδη τα οποία εισάγονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αλληλείς μας πρέπει να τηρούν μια σειρά προτύπων διοικητικών, ε, τεχνικών και προτύπων ελέγχου και πολλές φορές υποσκάπτονται από φθηνότερα και πολλές φορές κατώτερα προϊόντα τα οποία εισάγονται πολύ συχνά χωρίς κανένα προορισμό σε πολύ χαμηλές τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιούνται λοιπόν οι αλληλείς μα, γιατί δεν υπόκειται και τα εισαγόμενα προϊόντα στο ίδια πρότυπα που υπάγονται και τα δικά μας προϊόντα. Και επίσης αυτές οι εισαγωγές γιατί δεν υπάγονται στις ελάχιστες τιμές οι οποίες ε, ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονό ότι γενικά υπάρχει έλλειψη τέτοιων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, σε πολλές περιπτώσεις ε, τέτοια προϊόντα εχθείων ε, ε, αφαιρούνται από την αγορά γιατί δεν τηρούνται οι ελάχιστες επίσημες τιμέ. Για παράδειγμα πρόσφατα ε, τέτοια είδη υποκατάστατα, όπως τα ονομάζουμε, έχουν υπονομεύσει την παραγωγή των ε, Ευρωπαίων αλλιέων. Και ίσως ε, οι καταναλωτές να δίνουν και λιγότερη προσοχή στην ποιότητα και στην ανεχνησιμότητα των προϊόντων όταν βρισκόμαστε σε φάση οικονομικής ύφεση. Είναι όμως σωστό και δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέπει τέτοια προϊόντα τα οποία δεν τα ελέγχει σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των περιβάλλων, τις κοινωνικονομικές τους ε, συνέπειες. Είναι σωστό να επιτρέπεται να διστρεβλώνουν αυτά τα προϊόντα την, ε, τον ανταγωνισμό ως παραγωγή. Αναγνωρίζουμε ότι η βιώσιμη παραγωγή των ε, άγριων νυχτίων θα πρέπει να αποτελεί τον σκοπό μας. Και ενώ η παίζει σημαντικό ρόλο, δεν θα πρέπει να την επιτρέψουμε να στρεβλώσει τα τοπικά περιβάλλοντα και να αποσταθεροποιήσει τι αγορέ. Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί περιορατικοί όροι και ελάχιστε τιμέ για όλα τα εισαγόμενα ψάρια και ο καταναλωτή θα πρέπει να συνειδητοποιεί ακριβώ τι αγοράζει και τι σημαίνει η ποιότητα, η θρεπτική αξία, ο περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προϊόντο. Και θα πρέπει τελικά αυτοί να αποφασίζουν αν προτιμούν ε, νοπό, ψάρι, άγριο ψάρι, άγριες εκτροφή ή εκτροφής, ε, ψάρι εκτροφής ε, ή υδατοκαλλιέργειας. Θα πρέπει οι οργανώσεις ε, παραγωγών δικτύων να ενισχυθούν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Δεν θα πρέπει να καταργηθούν φυσικά οι ελάχιστες τιμές, αλλά θα πρέπει να αποτυπώνουν καλύτερα τις τοπικές ε, συνθήκες σε ό,τι αφορά τη διάθεση στην αγορά και θα πρέπει να γίνει μια απόπειρα να ενισχύσουμε και να οργανώσουμε τις τιμές σε περιφερειακό επίπεδο ή ένα λιμάνι. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει καλή κοιλία οργάνωση για τους πόρους της αγοράς αυτής. Η ανοιχνησιμότητα των πόρων είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντική. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς όρους των οργανώσεων ε, παραγωγών για την διαχείριση των αγορών και για την συνέχιση της βελτίωσης της οργάνωσης των προμηθειών. Μια ευρωπαϊκή ετικέτα η οποία θα καταδεικνύει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους ε, που ορίζονται στους τρεις πυλώνες της ΚΑΠ, οικονομία, κοινωνικά θέματα και περιβάλλον, αποτελεί μια σωστή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να ακολουθούμε τους εξής στόχους, να προσπαθούμε να βρούμε μια ε, ισορροπία σε ό,τι αφορά την προμήθεια και την ε, ζήτηση για να μεγιστοποιήσουμε την τιμή, να, σταθεροποιήσουμε τις τιμές και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του κοινωτικού στόλου. Η συνεργασία με τις οργανώσεις παραγωγών είναι κρίσιμη για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να περιληφθεί στη νέα ΚΑΠ προκειμένου να δώσει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθορισμός ε, τιμών προσανατολισμού, αν θέλετε, και αναφοράς και του μηχανισμού παρέμβασης θα πρέπει να παραμένουν ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, κοινή οργάνωσης αγοράς και οι μηχανισμοί αγοράς θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της πλήρους αποζημίωσης για το κόστος που προκύπτει και τις δίκαιες ανταμοιβή για τη δουλειά που γίνεται. Η πιστοποίηση και η, η ενίσχυση μάλλον και η υποστήριξη σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση και την ετικετοθεσία θα πρέπει να οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο για να μην υπάρχει δυνατότητα να απολούνται ψάρια εκτός των ενώσεων παραγωγών και προκειμένου να είναι και διαφανής και ανοιχτή η αγορά. Συνοπτικά θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε κατά πόσο θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι αλληλείς, που θεωρώ ότι είναι οι αλληλείς που υπόκεινται στην πιο υψηλή ρύθμιση στον κόσμο, να σας ρωτήσω λοιπόν αν, θεωρείτε ότι, αν πιστεύετε ότι αξίζουν να βλέπουν το ίδιο τους το την ίδια δουλειά να υπονομεύεται από τις ξένες εισαγωγέ. Θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθεί να έχει βιώσιμη αλληλεία σε 10 χρόνια. Το μόνο που ζητάμε είναι να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να ανταγωνιζόμαστε σε, με ίσους όρους. Ε, νομίζω ότι θέσατε κάποια ερωτήματα πολύ κέρια που αφορούν τις εισαγωγές και το θέμα της σήμανσης βεβαίως. Στη συνέχεια λοιπόν, για να αλλάξουμε κάπως τη σειρά. Είχαμε ε, προβλέψει δύο τμήματα στη συζήτηση με εκπρόσωπο ε, των ε, αλλιέων και εκπρόσωπο των μεταποιητών. Τώρα να δώσω, τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλερ που είναι εκπρόσωπος των μεταποιητών. Κύριε Κέλλερ, μπορείτε τώρα. Όπω συνήθω, αλλάζουμε όλο το πρόγραμμα, ολόκληρο το πρόγραμμα. Ε, τι να κάνουμε τώρα, άλλα προβλέπουμε. Κύριε Πισόν, για ελάτε. Βλέπετε ότι είμαστε πολύ ευέλικτοι. Ο κύριο Πισόν έχει το λόγο για 15 λεπτά. ça, oui. Bon, here <laughs> bon, je vais essayer d'aller vite, parce que j'ai compris. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα. Γιατί κατάλαβα, Πρόεδρε, όχι, όχι, πρόεδρο. Έχετε 15 λεπτά. Μην ανησυχείτε. Ε, θα σεβαστούμε το χρόνο που έχουμε προβλέψει για εσά. Δεν πρόκειται να σα κόψουμε το λόγο. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι ευρύτατο, και έχουμε εκπροσώπου των παραγωγών. Εγώ σκέφτηκα να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο αφορά ε, την ε, ε, επίδραση των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά. Βεβαίω αυτό σημαίνει δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα σημεία τα οποία ακούσαμε ήδη και τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ε, οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για μία σειρά από θέματα, ικανότητα παρέμβαση κτλ. Θα επικεντρώσαμε στην προσοχή μου στο συγκεκριμένο θέμα. Πρώτα απ' όλα να σα παρουσιάσω πολύ σύντομα την οργάνωσή μου. Είμαστε, έχουμε την έδρα μα στη Βρετάνη, στη Γαλλία. 562 ε, πλοία έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε τρία χρόνια χάσαμε περίπου το 30% της ελληνικής ικανότητας στην περιοχή αυτή. Ε, λόγω της ε, διαδοχικής εφαρμογής ε, σχεδίων εξόδου από την αλληλευτική δραστηριότητα για να είμαστε σύμφωνοι με την κοινή αλληλευτική πολιτική που μας ζητά να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην ικανότητα αλλήλευσης και στην αλληλευτική ικανότητα. Σήμερα έχουμε 74.000 τόνους λευκών ψαριών, πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό σε εθνικό επίπεδο. Είναι το 1 τρίτο της συνοπής αλίας στη Γαλλία, αλλά ε, θα καταλάβουμε στη συνέχεια ότι αυτά όλα είναι πολύ λίγα, λαμβάνοντα υπόψη ανάγκε τη ε, ευρωπαϊκή αγορά. Αν, αν εξετάσουμε τώρα τις μέσες τιμές των προϊόντων ε, που εκφορτώνουν τα μέλη μας, βλέπουμε την εξέλιξη των τιμών από το 2005 σε ευρώ και βλέπουμε ότι ότι μειώθηκαν οι τιμές μας, οι μέσες τιμές κατά 18% από το 2005 και ε, ε, ε, από το 2006 ιδιαίτερα έχουμε όξιση του φαινομένου αυτό, πολύ σημαντική, αυτού του, πολύ σημαντική μείωση. Πάντως αυτή η τάση παρουσιάζει διαφοροποίηση ανάλογα με τα προϊόντα. Έχουμε προϊόντα υποκατάστασης, Ε, τα, τα λευκά ψάρια και τα φιλέτα ψαριών ε, ε όσον αφορά το το μερλούκιο, ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μείον 48% από το 2006 μέχρι το 2009. Βλέπετε τι διακύμανση έχουμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό ε, και λόγοι που έχουν να κάνουν με την Αλία γενικότερα και, με τη, και ειδικότερα στην Βρετάνη. Βέβαια, η οικονομική κρίση που έχει επίπτωση στην κατανάλωση, και ε, επομένως και στις τιμές ε, που πολλούν τα μέλη μας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, γιατί αν ε, λάβουμε υπόψη και εξετάσουμε την εξέλιξη των τιμών σε άλλα είδη, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, ε, να πάρουμε, ε, για παράδειγμα, ορισμένα ψάρια όπως την πεσκανδρίτσα, ε, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν υποκατάσταση. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για αύξηση. Όσον αφορά το λαβράκι, για παράδειγμα, δεν, θα, δεν, θα, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά σχετικά πρέπει να σας πω ότι είμαστε αντιπροσωπευτικοί. Για την Πεσκανδρίτσα, για παράδειγμα, η οργάνωσή μου έχει 9.000 τόνους ε, ε, παραγωγής το χρόνο. Άρα στο 25% βρισκόμαστε του συνόλου της παραγωγής ε, πεσκανδρίτσας του Ατλαντικού. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιλώ γενικά για τις εκφορτώσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για ποια τάση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και εδώ θα ήθελα να μιλήσω στο σύνολο των προϊόντων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι οι ανάγκε είναι μεγάλες. Γιατί αν δούμε την ευρωπαϊκή αγορά θα δούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε κατανάλωση 13 εκατομμυρίων ε, ε, προϊόντος ισοδύναμου ζωντανού βάρους. Και αυτό συγκρίνεται το με τις 74.000 τόνους που παράγουμε εμείς. Βεβαίως ε, δεν τίθεται ζήτημα για μας ε, να αμφισβητήσουμε αυτή την ιδέα ότι δηλαδή απαιτείται, ε, απαιτούνται οι Βεβαίω δεν θέλουμε να αρνηθούμε κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ τα πράγματα πρέπει να τα δούμε ε, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή παραγωγή όλων των ειδών και τις εισαγωγές όλων των ειδών. Εδώ αν κάνουμε ε, αυτή τη σύγκριση θα δούμε ότι το 60% προέρχεται από τις εισαγωγές και το 40% από τις κοινωτικές εισαγωγές. Ε, Πρέπει επίσης να δούμε ότι ανάλογα με το είδος του προϊόντος ε, αυτή η διαφορά ε, ε, είναι, αλλάζει. Εάν δούμε τα λευκά ψάρια, για παράδειγμα, για τα οποία η κρίση της αγοράς είναι αρκετά σημαντική και την περιέγραψα και πριν από λίγο, και εδώ έχουμε ομαδοποίηση όλων των, ε, ε, των, των ψαριών του στυλ Μερλούκιος, Γάδος, ε, ε, ε Εγκλεφίνος, ε, Σολομός και τα παράδειγμα, και παράδειγμα συγγνώμη και τα λοιπά, θα δούμε ότι η εξάρτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. εδώ πλησιάζουμε ιδιαίτερα το 90% εξάρτηση από τα εισαγόμενα και 10% στήριξη στην κοινοτική παραγωγή. Και αυτό είναι σημαντικό που είναι σημαντικό να δούμε είναι ότι μειώνεται η παραγωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αυξάνονται οι εισαγωγέ. Και γιατί μειώνεται η παραγωγή. Λόγω τη απορρίθμιση που οδήγησε ε, σε μείωση τη αλληλευτική ικανότητα, μείωση των ε, δραστηριοτήτων ε, των αλληλευτικών, των σκαφών, σχέδιο διαχείριση του μπακαλιάρου κτλ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν 673.000 τόνους από το 2005 Δηλαδή, δύο φορέ η κοινωνική παραγωγή είναι η αύξηση αυτή. Βλέπετε λοιπόν γιατί μεγέθη μιλάμε. Ε, θεαματικά. Όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, δηλαδή εκτός των λευκών ψαριών, θα δούμε ότι και εδώ οι σχέσεις δεν είναι ίδιες. Δεν βρισκόμαστε στο 50-50, αλλά δεν απέχουμε και πολύ. 55% ε, είναι οι εισαγωγές σε σχέση με την ε, παραγωγή με την κατανάλωση μάλλον, και 45% ε, η κοινοτική παραγωγή. Τώρα, ε, παρά ε, αυτή την, την υψηλή ζήτηση και τις μειώσεις των τοπικών τιμών, όπως σας είπα και πριν από λίγο για τα λευκά ψάρια, εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ελευτική δραστηριότητα που οδεύει στη βιομηχανία. Και εδώ να σας δώσω του αριθμού τη οργάνωσή μου. Παράδοξο είναι ότι έχουμε μείωση των τιμών που φαίνεται με την μπλε αυτή καμπύλη, διορθώνει ο μιλητής, όχι, ναι, με την μπλε καμπύλη και την τάση με το κόκκινο βέλος. Και, και μία σχετική ε, αύξηση, ε, όπως βλέπετε από το ιστόγραμμα. Ε, sur, ε, sur le Merlu, on atteint maintenant 500 ε, tonnes de retraite βλέπετε ακριβώ τα στοιχεία ε, και το, και το τι ακριβώ γίνεται, λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί λοιπόν παρά τη μείωση αυτή εξακολουθούμε να έχουμε ε, αυτές τις ε, ε, αποσύρσεις. Αναφέρθηκε πριν από λίγο. Οι κοινοτικοί παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στις, στις τιμές. Γιατί ακριβώς ε, οι συμβάσεις δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις, ε, τα φαινόμενα αυτά των αποσύρσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις τρίτες χώρες. Και όταν δούμε τα είδη για τα οποία ο ανταγωνισμό ε, από τι τρίτε χώρε δεν είναι τόσο σημαντικό και αναφέρω την Πεσκανδρίτσα, εδώ όχι μόνο οι τιμέ είναι σταθερέ, αλλά και οι αποσύρσει είναι αμεληταίε. Παράδειγμα, αυτό που σημειώθηκε το 2009 ήταν 3 τόνοι, ενώ είχαμε νέα τόνους παραγωγής. Βλέπουμε λοιπόν ε, με αρκετή σαφήνεια ότι η πίεση εκ των έξω, των προϊόντων δηλαδή που εισάγονται ε, στην ιστορική αγορά, είναι, γίνεται αισθητή σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και στην ουσία η Ευρωπαίοι παραγωγή ε, δεν είναι, μπορούμε να το πούμε. Αλλά γιατί δεν είναι κατά την άποψή μου, μία από τις εξηγήσει για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ε, παραγωγών και μάλιστα να σας πω ότι τα στοιχεία που δίνω εγώ εδώ ε, ε, προέρχονται από στοιχεία 2004, στοιχεία του ΦΑΟ, αλλά εδώ έχουμε κάποια στοιχεία για να δούμε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και δραστηριότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ παίρνω στοιχεία για ανάλογα πλοία, εδώ για βενθοπελαγικές στράτες. Κοιτάξτε λοιπόν τι κοστίζει ένας ναυτικός αναημέρα στη θάλασσα. Στα αριστερά βλέπετε ότι στη Γερμανία ή στη Γαλλία χοντρικά ε, ένας ναυτικός σε μία ε, τράτα 20 μέτρων ε, κοστίζει 160 δολάρια και κοστίζει το ίδιο άτομο 22 δολάρια στην Σενεγάλη. Και σε μία έκθεση της ε, αρμόδιας γενικής διεύθυνσης ε, που ε, αναφέρεται στο σύστημα των γενικευμένων προατιμήσεων και που αναφέρει ότι εδώ θα πρέπει να συνδυάσουμε τις πολιτικές ανάπτυξης αλλά να δούμε τι γίνεται και τι γίνεται με την εξάλληψη της φτώχειας και την πρόθεση της αηφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Δηλαδή, επιτρέποντας και προωθώντα το εμπόριο με βάση αυτό το επίπεδο ανταγωνιστικότητα, εξαλείφουμε τη φτώχεια στι χώρε αυτέ. Ε, θέτω απλά για μόνο το ερώτημα, κοιτάξτε τα στοιχεία και δεν έχω απάντηση. αν λοιπόν ε, πάμε παραπέρα και θέλουμε να δούμε τις επιπτώσεις αυτής της ε, διαφοράς του κόστους στη ε, σε σχέση με την εκμετάλλευση των πλοίων, βλέπετε τι γίνεται συνέχεια. Εδώ έχετε ε, τον κύκλο εργασιών των πλοίων ε, και το μερίδιο ε, των μισθών. Στη Γερμανία πέραν του 40% του κύκλου εργασιών χρησιμοποιείται για τις πληρωμές, για τους μισθούς, για, την, για το πλήρωμα. Ενώ είναι λίγο περισσότερο από 15% το ίδιο ποσοστό στη Σενεγάλη, στην Αργεντινή, στην Νότια Αφρική. Υπό αυτές τις συνθήκες Μάλιστα, μπορεί κανεί να μειώσει τις τιμές και να είναι ανταγωνιστικός στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, και να ρίχνει τις τιμές με τον τρόπο αυτό. Μα ακριβώς γι' αυτό εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί στην ε, αγορά των λευκών ψαριών ε, μέσα στα δικά μας τα σύνορα. Και βεβαίως δεν έχουμε την ικανότητα να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί γιατί ο στόχος ε, των Γάλλων κυρίων πλειοκτητών δεν είναι ε, να ε, απασχολούν ανθρώπους που τους πληρώνουν, πληρώνουν 22 δολάρια, μα δεν είναι αυτή η αναπτυξιακή πολιτική. ούτε θα προωθήσουμε την οικονομία στις ακτές της Ευρώπης, ούτε όμως και την ανάπτυξη σε Νεγάλη στην Αργεντινή. Υπό αυτές τις συνθήκες, για να δούμε λίγο το μέλλον των πλειοκτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το θέμα τη ανταγωνιστικότητα που έχει να κάνει με τη διαφορά ε, του κόστου του εργατικού δυναμικού. Έχουμε βεβαίω και άρση ε, βαθμιαία των τελωνιακών φραγμών με βάση του κανόνε ε, του ΠΟΕ και βεβαίω και με τι επιθυμίε της Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει ε, τις πόρτες της ε, στις εισαγωγές. Επίσης, ε, μείωση των επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν ε, οι δεσμεύσεις του Johannesburg. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλα τα συμβαλώμενα μέρη, αποφάσισαν από το 2015 το σύνολο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με βάση την αηφόρο διαχείριση. Αλλά δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε τις δεσμεύσεις αυτές και οι υπόλοιποι. Ε, αυτό για μας κάτι σημαίνει. Αυτή η μείωση των επενδύσεων που έχει να κάνει με την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης με στόχο την αηφορία, δηλαδή μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης, ε, αντιμετώπιση των αποθεμάτων, μείωση του αριθμού των ε, πλοίων κτλ. Μα όλα αυτά θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη μείωση της κοινωνικής παραγωγής. Και βλέπουμε ήδη τις επιπτώσεις, γιατί το μερίδιο της κοινοτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται όλο και περισσότερο λόγω αυτής της πίεσης από τις χαμηλότερες τιμές των εισαγόμενων προϊόντων που φτάνουν χωρίς τους ίδιους περιορισμούς όμως γιατί δεν έχουν αντιμετωπίσει τέτοια βάρη η παραγωγή αυτή. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη ε, δυσκολία και αποδυνάμωση της παραγωγής στην Ευρώπη. Προσανατολισμοί, τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να απαιτήσουμε την, ε, ε την ε, συμμόρφωση όλων με τις δεσμεύσεις του Johannesburg. Εμείς ε, προσπαθούμε να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αηφόρο διαχείριση των αποθεμάτων μας, αλλά και, και με αυτόν τον τρόπο πληρώνοντας όλες τις θυσίες ε, και πληρώνοντας το τίμημα, ε, αλλά οι υπόλοιποι ξεχνούν τις δεσμεύσεις του Johannesburg. Όπως μπορέσαμε λοιπόν να επιβάλλουμε και, τους, ε, ε, και τα ε, υγειονομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες που κάνουν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και όσον αφορά τα αλληλευτικά πρότυπα. Έτσι ώστε και οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι 2015 όλα όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται θα αποτελούν αντικείμενο διαχείριση με βάση του κανόνε αυτού, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρε που κάνουν εξαγωγέ ε, έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια με αξιόπιστα μέσα για να οδηγηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Τώρα μια λεπτομέρεια. Είναι παράλογο από τη μια να έχουμε μείωση παραγωγή μείωση των τιμών, ε, αύξηση της απόσυρσης. Και αυτό δεν ε, οφείλεται μόνο ε, στους μεταποιητές της Ευρώπης, γιατί υπήρξε μια στιγμή όπου η παραγωγή μας μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο χρησιμοποίησης από τους μεταποιητές και όμως δεν τη χρησιμοποιούσαν. Γιατί, γιατί ε, το σύστημα στήριξης της ε, αγορά στην Ευρώπη δεν είναι προσαρμοσμένο, δεν είναι επικαιροποιημένο, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν ε, οι τιμέ απόσυρση, παρέμβαση κτλ. Είναι τεχνικά όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικά. Και τέλος, τελειώνω, γιατί ήδη βλέπω ότι ξεπέρασα το χρόνο μου. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο ότι στην τελευταία ανάλυση ο καταναλωτής να ξέρει τι ακριβώς καταναλώνει. Όχι μόνο λοιπόν να γνωρίζει την προέλευση του προϊόντος που αγοράζει, αλλά ε, πού έγινε η πρώτη μεταποίηση. Και αυτό είναι ουσιώδης σημασία και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με ε, τον άνθρακα, ε, τι, τι γίνεται δηλαδή από άποψη εκπομπών και ε, τι γίνεται με τις δεσμεύσεις του Ιωάννησμπουργκ, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ζητώ συγγνώμη τη μακρηγόρησα. Eh, Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και τα θέματα που θέσατε. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μια συζήτηση 45 λεπτών. Ο κύριος Βαλές έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο δεύτερο τμήμα ήθελα να θέσω την ε, ερώτησή μου, να απαντήσω όμως ε, σε κάτι που είπε ο κύριος Στίβενσον για την ανιχνευσιμότητα των ε, αλλιευτικών ειδών. Προφανώς υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει χαμηλή δυνατότητα ανέχνευσης, αλλά σύμφωνα με, τον, με τους κοινωνικούς αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Αν δείτε τα κατεψυγμένα προϊόντα, ή τα συσκευασμένα προϊόντα. Ε, βλέπετε ότι όταν ε, είμαστε στο Ιανεμπόριο υπάρχει πληροφορία για τη χώρα προέλευσης, αλλά το βασικό ζήτημα είναι η ποιότητα του ψαριού στα σούπερ μάρκετ. Το κατεψημένο ψάρι που πωλείται σε σούπερ μάρκετ δεν είναι νοπό πραγματικά. Και πολλές φορές δεν είναι και καλό. Να ρωτήσω λοιπόν τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Η το σύστημα ελέγχων της Ένωσης εγγυάται και σε τι βαθμό ότι τα αλληλευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση δεν αποτελούν κίνδυνο για τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, ένα ψάρια από την Άπο την Κίνα. Η παραγωγή εκεί τήρει τις απαιτήσει που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Merci, Madame la euh, euh, ευχαριστώ πρόεδρε. Να υπογραμμίζω καταρχάς ότι οι τρει ε, ομιλητές που προέρχονται από οργανώσει παραγωγών βεβαίω ανέφεραν και οι τρει τα τρία προβλήματα, τα ίδια προβλήματα που προέρχονται από τι εισαγωγέ από τρίτε χώρε. Μιλάμε για ανιχνευσιμότητα, για μακροχρόνια μακροχρόνια θέμητο ανταγωνισμό έναντι των Ευρωπαίων αλλιέων, είτε είναι από τη Σκωτία, είτε είναι από τη Γαλλία, είτε από την ε, Ισπανία. Και θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές ε, αργότερα. Καταλάβαμε ωστόσο αυτή τη στιγμή ότι όλοι έθεταν τα ίδια ζητήματα και ανέφεραν τα ίδια προβλήματα. Προφανώς σε ορισμένα είδη, το ανέφερε ο κύριος Πίσω, για τα οποία υπάρχει μικρός ανταγωνισμός με είδη που προέρχονται για παράδειγμα από την από υπάρχουν ε, λιγότερα προβλήματα. Το λαβράκι π.χ. Άλλα προϊόντα που μοιάζουν με κοινοτικά δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Οι εισαγωγέ δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Μας δείξετε και ένα γράφημα που δείχνει το κόστος ε, της εργασίας. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον γράφημα, το είχαμε συζητήσει και στο κείμενό μας, πρέπει να το δούμε. Βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των 160 δολαρίων. Δολάρια λέτε εδώ, καλύτερα θα να λέμε εμείς ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Όταν στη Γερμανία το κόστος είναι 160 και στη Σενεγάλη 20 δολάρια, καταλαβαίνουμε την τεράστια διαφορά. Εγώ πάντως Πιστεύω ότι και οι τρεις ομιλητές έφεσαν πολύ σωστά το πρόβλημα που εξετάσαμε ήδη στο κείμενο εργασία που έχουμε μπροστά μας. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν συμβολή που ελπίζω να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Λοβίν. Ευχαριστώ τους ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή τους. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση του Σκοτσέζου ομιλητή, κάτι που επανέλαβε και ο Γάλλος. Η ελάχιστη τιμή για τα ψάρια και η αποφυγή μείωσης τιμής μέσω της ε, απόσυρσης κάποιων ειδών. Εμείς πρέπει να δούμε την κατάσταση για να προστατεύσουμε προφανώς τους αλληλείς μας, αλλά να μην, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε μια στρεβλή κατάσταση που συνέβη στο παρελθόν και συμβαίνει και τώρα για τις γαρίδες στην Σουηδία. όπου το προϊόν προσπαθεί, ε, όπου το προϊόν για να μείνει σε υψηλή τιμή, ε, αποσύρεται. Δηλαδή, μπαίνουν τα συστήματα απόστησης, ε, αυτό έχει γίνει στο παρελθόν στην Σουηδία, που οδήγησε στην χώρα να μην χρησιμοποιηθούν 5.000 τόνοι προϊόντος ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς όπως ε, ζωοτροφές δυσκολεύοντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του προϊόντος σε μεταγενέστερη φάση μέσω της κατάψυξης για παράδειγμα. Τελικά το προϊόν καταστράφηκε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση όπου όχι μόνο υπάρχει πίεση στην, ε, στο απόθεμα αλλά και έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευρά καταναλωτών. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη Σουηδία και είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση. Στην ουσία δηλαδή οι Σουηδοί δεν ε, ψαρεύουν για τα μαγαζιά, ψαρεύουν για την απόσυρση. Αυτό έχει αρνητικέ συνέπειε και για τον κλάδο και θα ανακούσω τι απόψει των εκπροσώπων. Κύριε Πρεσβάρια. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, ομιλητές. Ε, νομίζω ότι μιλήσατε πολύ σωστά για τα προβλήματα αυτά και για τα, όπως είπε ο κ. Καντέκα, αυτά που αφορούν την αγορά πολύ σημαντικά. Θέσατε το θέμα των εισαγωγών, των μισθών, της εμπορίας. Κύριε Στίβενσον, θέσατε ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε κάπω. Μιλήσατε για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην οποία αλία και στην υδατοκαλλιέργεια, στην ιστιοκαλλιέργεια. Μα νομίζω ότι και η ιστιοκαλλιέργεια αποτελεί τμήμα τη αλίας. Τουλάχιστον ε, αυτό θα πρέπει να γίνεται. Αποτελεί μέρο τη αλληλευτικής πολιτική και μέρος τη λύση. Τώρα, τέθησαν δύο ζητήματα σε σχέση με τι πιθανέ λύσει. Ο τελευταίο ομιλητής μίλησε για πρόβλημα εμπορία και το συνέβησε με του μισθού. Μια πιθανότητα θα μπορούσε να είναι ε, το βασικό ε, εισόδημα των αλλιέων. Και επίση ακούσαμε ω πιθανή λύση την εξατομίκευση των επιχειρήσεων. Μπορείτε να μα εξηγήσετε πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει ε, προ την κατεύθυνση εξέβρεση τη λύση. Η κυρία Ρόντου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και του τρει ομιλητέ πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε. Ωστόσο, ένα πρόβλημα με απασχολεί και στους τρεις ομιλητές ε, άκουσα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές μεγάλη κριτική. Αλλά σε ό,τι αφορά την βετοκαλλιέργεια και πάλι διστακτική είναι. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του συναδέλφου Κίντο Μιλάνα η οποία υποδεικνύει ότι η διδοκαλλιέργεια στην Ευρώπη βρίσκεται σε πρώιμη φάση ακόμα και σε σύγκριση με άλλες χώρες θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω. Εσείς, ως ε, οργανώσεις παραγωγών, αν ε, τοποθετήσετε τόσο επικριτικά Θεωρώ ότι αυτό παρουσιάζει προβλήματα για την συνολική αλληλευτική πολιτική της ε, Ένωσης. Και ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω για την ε, πιστοποίηση. Στην Γεωργία προτείνουμε από τη γέννηση ενός ζώου μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά ε, ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας, πιστοποίησης. Αυτή η πιστοποίηση δεν είναι ενδιαφέρουσα και για εσά. Δηλαδή από την πρώτη φάση μέχρι τη διάθεση της αγοράς να υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίηση. και αν ε, προάγατε την πρακτική αυτή από συνεργασία μαζί μας δεν θα πείθαμε με τον τρόπο αυτό τον καταναλωτή να αγοράσει ποιοτικά υψηλότερα προϊόντα και νομίζω ότι έτσι λοιπόν δεν θα προωθούσαμε και την ευρωπαϊκή αγορά σε σύγκριση με τι ξένε αγορέ. Ευχαριστώ κύριε Σάντη Πεσέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές για την ε, συμβολή του κύριου Τεϊσέιρα, ο οποίος αναφέρθηκε στη στο σημαντικό ρόλο που παίζουν οι οργανώσει των παραγωγών. Εδώ πρόκειται όμω για το εξή ερώτημα. Οι αλληλεί. ε, το μερίδιο των αλλιέων, αν θέλετε, στην τελική τιμή πώληση. Ε, και τι γίνεται με την ποιότητα. Ε, δίνεται το βάρος που θα έπρεπε στην ποιότητα και ε, στις σχέσεις με, τους, ε, με, τις, ε, με τα διάφορα, με τις διάφορες οργανώσεις διανομής. Κύριε Στίβενσον, αυτό που είπατε και που μου τράβηξε την προσοχή είναι ε, τι ελάχιστε τιμέ σε σχέση με συγκεκριμένα είδη. Μα αυτό που λέτε δεν μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και όσον αφορά τον κύριο Πισόν, που μίλησε για τα αλληλευτικά πρότυπα, μήπω μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερα για το σημείο αυτό. Τι πιστε, ποια πιστεύω θα μπορούσαν τα πρότυπα αυτά. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια. Πρώτο σχόλιο. Ε, σε σχέση με την ε, κοινή ελευτική πολιτική. Η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ ε, έχει αναφέρει ορισμένε ιδέε που έχουν να κάνουν και με τα σχέδια ανάκτηση, ε, όπω για παράδειγμα το Μερλούκιο του Βορρά Δηλαδή ότι αν μειώνεται η ελευτική δραστηριότητα τότε θα αυξούν οι τιμές. Αυτό ήταν η ιδέα, μα βλέπουμε ότι αυτός ο κανόνας στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Ο κύριος Πισόν μάλιστα το είπε σαφώς ότι ανάλογα με τα είδη υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες διαφορές. Ε, και όσον αφορά το Μερλούκιο, θέμα το οποίο έχω μελετήσει και εγώ, τα αποθέματα του Μερλούκιου του Βορρά, στο οποίο αναφέρθηκε ε, ο κύριο Πισόν και στη δική μου την περιοχή, στη Γαλλικία. Η τιμή είναι ακριβώ η ίδια εδώ και πολλά χρόνια. Α, το αν μειώνεται η αλία, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται οι τιμέ. Ε, εντάξει, βεβαίω όταν αλλιεύσει κανεί υπερβολικά και ρίξει όλο το προϊόν στην αγορά θα πέσουν οι τιμέ, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Και το παράδειγμα αυτό που σα έδωσα είναι σαφέ. Γιατί το, το ψάρι αυτό έχει υποκατάστατα ε, άλλα είδη μερλούκι, όπω για παράδειγμα αυτά που έρχονται από, το, από τη Νότια Αφρική ε, ή ο παγκάσιο που έρχεται από το Βιετνάμ. Όλα αυτά λοιπόν τι σημαίνουν. Ότι έρχονται υποκατάστατα στην αγορά και πλήττεται με αυτόν τον τρόπο ένα τομέα που επιπλέον έχει κάνει και την προσπάθεια για μείωση τη ελληνική δραστηριότητα και δεν βλέπει ε, αύξηση των εισοδημάτων του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η ιδέα που πάντα αναφέρεται στι αναλύσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τα ε, σχέδια ανάκτηση και διαχείριση είναι λανθασμένη. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει εν ώψη τη μεταρρύθμιση τη αλληλευτική πολιτική, έτσι ώστε να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένε προτάσει ε, και πιο ρεαλιστικέ. Και κάτι άλλο που θα ήθελα επίση να αναφέρω είναι το εξή και να ρωτήσω ε, και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Και εδώ ο κύριο Πισόν είπε κάτι σαφέστατο. Όχι μόνο αυτή η εμπορική πολιτική που είναι τελείως αποδεσμευμένη από τα συμφέροντα των αλλιέων και θα κάνουμε την ε, ε, ερώτηση συνέχεια στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Ε, και, και όχι μόνο σήμερα, αλλά και, και τις προάλλες συζητήσαμε το θέμα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο πραγματικά εξαλείφουμε τη φτώχεια στις χώρες αυτές. Και ακούσαμε και σε προηγούμενη συνεδρίαση ένα παράδειγμα από τη βιομηχανία στη χώρα των Βάσκων. 260 δολάρια παίρνει ένας υπάλληλος ε, που εργάζεται στη βιτική βιομηχανία στη Γαλλικία και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ για παράδειγμα, όχι, όχι, όχι στο Βιετνάμ, στην Ταϊλάνδη, στην Ταϊλάνδη ήταν το παράδειγμα, λέει η πρόεδρο. 60 δολάρια θα έπαιρνε ο άνθρωπο αυτό. Και μάλιστα έκαναν εισαγωγή εντό εισαγωγικών σκλάβου από τη Βυρμανία που έπαιρναν 40 δολάρια. Καταλαβαίνετε ε, τι γίνεται δηλαδή με την παππούα και με τη Νέα Γουινέα αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε για τους κα, ε, κανόνες καταγωγής και κάποιος θα μιλήσει στο θέμα αυτό από τους ομιλητές. Ο τομέας ε, στην παππούα Γουινέα ε, αντιμετωπίζει φαινόμενα απεικιοκρατίας από την Ταϊλάνδη. Δηλαδή, όχι μόνο παίρνουν λιγότερα, αλλά αντιμετωπίζουν και τέτοια φαινόμενα και τέτοιε πρακτικέ. Ε, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν έχουμε εξάλληψη τη φτώχεια, αλλά προώθηση τη φτώχεια. Έχω μια ερώτηση λοιπόν προς τις δύο Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια είναι η σύνδεση που γίνεται όταν αποφασίζετε μια, και προωθείτε μία θέση, πώς εφαρμόζεται αλλού. Δηλαδή, ε, ε εμεί αποφασίζουμε κάτι για την Ελία, αποφασίζετε κάτι με, με την Ελία, σε επίπεδο Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Πώ συνδέεστε με τα εμπορικά θέματα όμω και με την εμπορική πολιτική. Γιατί ακούμε τι επικρίσει από όλου. Δεύτερον, αξιολόγηση αντικτύπου κάνετε ανάμεσα στις αποφάσεις που λαμβάνετε, οι υπουργοί εμπορίου αν θέλετε, ε, και τις, και επιπτώσεις ε, στην Ελία. Γιατί αυτό το οποίο είναι σαφέ αυτή τη στιγμή είναι ότι οι μαζικέ και ανεξέλεγκτε εισαγωγέ, και εδώ φταίνε τα κράτη-μέλη, έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε μεγάλο μέρο και τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά λοιπόν εκμηδενίζουν τις προσπάθειές μας και ε, τη βιομηχανία μας. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Όσον αφορά το θέμα ε, της, ε, ε της οικολογικής σήμανσης, πιστεύετε ότι κάποιοι σαφείς κανόνες προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να επιλύσουν εν μέρει ορισμένα από τα προβλήματα αυτά. Είναι μια ερώτηση που σας ε, απευθύνω. Εγώ δεν έχω την απάντηση. Έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι ε, έχω καταλάβει τι λέει ο, ο κλάδος όχι μόνο σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε επίπεδο και πιθανών εισαγωγών. Μήπως με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που αναφέρατε κι εσείς. Λοιπόν, να σας δώσω το λόγο. Πρώτα απ' όλα στην... Όχι, όχι. Ο κύριος Γκάλαγκερ που είχε σηκώσει το χέρι την τελευταία στιγμή. Πού είστε, εκεί. Ωραία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να κάνω και εγώ κάποια σχόλια η ακρόαση εδώ σήμερα το πρωί έχει εκπροσώπου από την Ισπανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και του καθεξή. Ουσιαστικά θα μπορούσαν οι ομιλητέ να είναι από οποιαδήποτε χώρα, γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα αλληλευτικά κράτη. Οι τιμέ του λευκού ψαριού και των ε, μαλακών σακών στην παρούσα φάση είναι ε, πολύ χαμηλέ και αγωνίζονται να επιβιώσουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και στα προηγούμενα, σε προηγούμενες θητείες και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μίλησαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά ζητήματα αυτά που ανακύπτουν, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για τους νέους αλληλείς και μάλιστα υπήρξε και ένα ευρύτερο σχέδιο, πρόγραμμα απόσυρσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι Παράλληλα με τη μείωση του στόλου θα υπάρχει ευρωπαϊκό ψάρι το οποίο θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά και ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των εκλογών. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα. Μας οδήγησε να πιστέψουμε ότι θα υπήρχε μια αναθεώρηση, μια κοινή οργάνωση της αγοράς από το 2011 και τώρα μας λένε ότι μπορεί η ημερομηνία αυτή να μετατεθεί στο 2014. Μα είναι ρεαλιστικό αυτό, να πάρει άλλα 3-4 χρόνια προτού ε, οριστούν οι νέοι κανόνες. Και τι θα κάνει η ελευτική, ο ελευτικός κλάδος. Ο κλάδος θα έπρεπε να είναι όπως οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί κλάδοι. Αλλά πώς υπέδειξαν και οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεβαίνει το κόστος και οι τιμές των ψαριών δεν αυξάνονται ανάλογα και άρα περιορίζονται διαρκώς τα περιθώρια και δεν υπάρχει ελκυστικότητα φυσικά στον κλάδο όσο για τις τράπεζες. Δεν είναι διτεθειμένες πλέον να αναλαμβάνουν κινδύνους. Πόσο λοιπόν θα γίνουν τέτοιες επενδύσεις αν δεν υπάρχει σιγουριά για το επίπεδο των τιμών για την πρώτη ο αλευτικός κλάδος παρεμποδίζεται από το εργατικό κόστος και δικαίως, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα λογικό εισόδημα, εύλογο εισόδημα και για τον παραγωγό και για τον μεταποιητή και για τις οικογένειες τις οποίες ε, πρέπει να υποστηρίξουν. Και δεν γίνεται με ίσους όρους ο ανταγωνισμό με τι εισαγωγέ από τρίτε χώρες. Είναι πραγματικά γελία η κατάσταση. Φυσικά και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν εισαγωγέ. Γιατί πρόκειται για ψάρι υψηλή πρωτεϊνικής αξίας, αλλά να γίνεται ανταγωνισμός με ίσους όρους και φυσικά να υπάρχει και μία ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να υπάρχει μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής και μία βασική σύσταση είναι ότι εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσουμε ό,τι πίεση μπορούμε για να επιταχύνουμε αυτή την μεταρρύθμιση της πολιτικής, γιατί τα πέντε χρόνια δεν είναι σωστό χρονικό διάστημα. Σε πέντε χρόνια θα έχει εξαλειφθεί η βιομηχανία, ο αλευτικός κλάδος που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πιο σημαντικός, αν θέλετε, για από άλλου κλάδους, γιατί παρέχει θέσεις απασχόλησης σε αποκεντρωμένες, εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και περιφέρειες της Ένωσης. Να μην περιμένουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα θα διορθωθεί από μόνο του. Δεν πρέπει να διορθωθεί από μόνο του. Πρέπει εμείς να αναλάβουμε δράση. Και όταν σκέφτομαι ότι το 2007 Μόνο 10 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν στο πρόγραμμα παρέμβασης. Ήταν τεράστιος προπολογισμό που είχαμε τότε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τις σχετικές οργανώσεις και θα πρέπει αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τους εκπροσώπους του κλάδου που βρίσκονται εδώ σήμερα, γιατί αυτοί κατανοούν πλήρως από πρακτικής άποψης το τι θα πρέπει να γίνει. Ο κύριος Φερέιρα, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δύο σύντομε παρατηρήσει για να υπογραμμίσω εκ νέου την ανάγκη που ανέφερε ο κύριος Γκάλαχερ, την ε, μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωση αγοράς. Το 2002 υπάρχει μία ανάγκη ε, μεταρρύθμισης της αγοράς. Βλέπουμε στο σημείο μου ότι e τα προϊόντα αυτά είχαν 0,16% των παρεμβάσεων μόνο. Το 20% του, της παραγωγής το 0, των οπών το 0,7 της αξίας ήταν το κέρδος αυτός. Έχουμε, έχουμε λοιπόν μια δυνατότητα πολύ περιορισμένης παρέμβασης σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Το περιγράψαν οι ομιλητές σήμερα. Πολύ λίγα εργαλεία της κοινή οργάνωσης εργολάς για επιθεώρηση, μικρή οικονομική δυνατότητα, αδυναμία της Επιτροπής να αναλάβει δράση, μετάθεση για μετά τις για μετά το 2012. Πρόκειται για θέματα σημαντικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η μεθοδολογία της εμπορίας. Οι τιμές είναι στάσιμες στο επίπεδο της παραγωγής, αλλά στον καταναλωτή δεν είναι. Αυτά τα στοιχεία ε, προκύπτουν από τις εισαγωγές προφανές που αλλοιώνουν με σημαντικό τρόπο την αγορά. Άρα πρέπει να δούμε και το πώς μπαίνει στο εμπόριο το προϊόν. Υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης αρκετά σημαντικές. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την υποστήριξη κατά άποψή μου των οργανώσεων των παραγωγών παρεμβαίνοντας στην η φάση της αλυσίδας παραγωγής. Αυτό είναι μια πιθανή λύση, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Γιατί οι οργανώσει των παραγωγών στην πλειοψηφία τους συγκεντρώνονται σε τρία κράτη μόνο. Άρα και εδώ ε, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης της Ευρώπης χρειάζονται και άλλα εργαλεία. Θα πρέπει να εξετάσουμε για παράδειγμα την δυνατότητα να υπάρχουν εγγυημένε τιμές ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους παραγωγούς. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, πρέπει να τη δούμε. Μέγιστο ποσοστό κέρδους. Αυτό επίσης είναι ένα εργαλείο που είχαν τα κράτη στη διάθεσή τους πριν τεθεί σε ισχύ η κοινή αλληλευτική πολιτική. Υπήρχε στην Πορτογαλία αυτό το μέγιστο ποσοστό κέρδους που επέτρεπε να αποτιμηθεί η τιμή στην πρώτη πώληση και να υπάρχει μια πιο δίκαιη ε, λειτουργία της αλυσίδας ε, της ε, αλυσίδας αγοράς. Αυτό με την κοινή αλευτική πολιτική χάθηκε. Τώρα, άλλα θέματα όπως πιστοποίηση, επισήμανση παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίλυση κάποιων από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Δεν είναι μία γενική παγκόσμια λύση, ούτε θα αποτελέσουν την πανάκια. Ωστόσο, η πιστοποίηση και η επισήμανση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν θα πρέπει να αποτελέσουν επιπλέον κόστος για τον παραγωγικό δεν μπορεί να είναι ένας παράγοντας στην αλυσίδα παραγωγής που θα κάνει ακόμα πιο άδικη την κατάσταση για τον παραγωγό. Πρέπει να υπάρχουν εγγύησεις ότι η πιστοποίηση θα προστατεύει τα συμφέροντα του κοινού και ότι κατά συνέπειο θα υπάρχει μία κρατική εγγύηση. Όχι όπως γίνεται τώρα η πιστοποίηση. Τώρα η πιστοποίηση είναι μια ακόμα ευκαιρία ε, εμποϊκής, εμπορικού κέρδους. Να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Επιτροπής και μετά θα λάβουν το λόγο καθένας από τους τρεις συγητές. Πρώτον, για την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, κύριε Γκαρθία Φεραίρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να διαπιστώσω καταρχάς ότι οι εισαγωγές συμφωνούμε όλοι, είναι αναγκαίες για να τροφοδοτηθεί η εσωτερική αγορά. Γιατί η κοινοτική αγορά δεν είναι επαρκής. Κατά 65% εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές. Επίσης, να σας αναφέρω μια μελέτη που είχε ξεκινήσει η Γενική Διεύθυνση Μάρια και που δημοσιεύτηκε πέρυσι. Το Μάιο του 2009 συγκεκριμένα. Αν δείτε τις αναλύσεις που περιλαμβάνει η μελέτη αυτή, εξέτασε πώς μπορούν να επηρεάσουν οι εισαγωγές τις τιμές ε, και την κοινωνική παραγωγή. Και το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι οι εισαγωγές δεν οδηγούν σε βλάβη της κοινωνικής παραγωγής, σε ζημία της κοινωνικής παραγωγής και ότι υπάρχουν εισαγωγές όταν είμαστε ικανοί να ικανοποιήσουμε την εσωτερική αγορά. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Επίσης, άλλο θέμα που περιλαμβάνει η έκθεση και θέλω να τονίσω είναι το εξής τα επόμενα έτη θα αυξηθούν οι εισαγωγές χωρίς να υπάρξει αρνητικός γενικός αντίκτυπος στην κοινωτική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζουμε ότι όπως αναφέρθηκε στην τελευταία συνέντευξη της Επιτροπής Αλληλείας από τον κ. η γενική τάση που υπάρχει θα συνεχιστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό σημαντική η μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, τόσο ώστε ο κλάδος να προσαρμοστεί και να είναι ανταγωνιστικός, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον ότι σε πολυμελές, σε πολυμερές επίπεδο θα υπάρξει μείωση των δασμών κατά πάση πιθανότητα, κάτι που είναι μια γενική τάση. Η αναπτυξιακή διάσταση που πολλοί ομιλητές ανέφεραν και η πρόεδρος μάλιστα, περιλαμβάνει τα εξή στοιχεία. Ε, τα τελευταία 40 χρόνια η αναπτυξιακή βοήθεια ήταν σημαντική και κάτι που οδήγησε σε αύξηση των ε, εισοδημάτων των χώρων αυτών λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους, της διαφοροποίησης οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίω στις γυναίκες, κάτι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά αυτό το level playing field που αναφέρθηκε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μια σειρά γεγονότων. Πρώτον, οι φυτοϊγειονομικές και υγειονομικές προϋποθέσεις της Ένωσης από τις υψηλότερες στον κόσμο πολλές φορές χαρακτηρίστηκαν ως προστατευτικές ρυθμίσεις αλλά είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η επισητιστική ασφάλεια του καταναλωτή. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι με τις απαιτήσει αυτές εξασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα που μπαίνουν στην κοινωτική αγορά τηρούν τις προϋποθέσεις και είναι ικανοποιητικές και ασφαλείς για τον καταναλωτή. Δεύτερον, υπάρχει ο κανονισμό κατά τη παράνομη ελεία που εξασφαλίζει επίση την ανεχρεσιμότητα των ε, προϊόντων. Η Γενική Διεύθυνση Trade μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Mare ενεπλάκει σημαντικά στην υλοποίηση και συνεργασία με τρίτε χώρε για να εξασφαλίσει ότι η θέση ισχύ του κανονισμού δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και θα εξασφαλίσει ότι οι εισαγωγέ θα προέρχονται από νόμιμε πηγέ και θα είναι και από βιώσιμη αλίευση. Τρίτον, κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα όταν διαπραγματεύεται η Επιτροπή Εμπορικέ Συμφωνίε, συμπεριλαμβάνει πάντα ένα κεφάλαιο που λέγεται Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων δεσμεύσει από πλευρά τρίτων χωρών ώστε να εφαρμόζουν ουσιαστικά τις συμβάσεις ε, του Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας και άλλων οργανισμών για, την, ε, για το περιβάλλον. Αυτό ε, ε, σημαίνει ότι ναι, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε δικά μας στάνταρντ, αλλά δεσμεύονται τα κράτη να τηρούν τα διεθνή στάνταρντ. Άλλο θέμα σημαντικό, κατά την άποψή μου, που θα ήθελα να υπογραμμίσω, και μιλώ για την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι για τον αντίκτυπο των ε, πολυμερών συμφωνιών στο εμπόριο, είναι ότι μόνο 5% των προϊόντων αλίας που μπαίνουν στην κοινωτική αγορά πληρώνουν, καταβάλουν το πλήρη δασμό, όπως τον αποκαλούμε. Το... Ένα μεγάλο ποσοστό μπαίνει είτε χωρίς δασμό, είτε με δασμολογική αναστολή, ενώ το 50% μπαίνει με, ε, προτι... με δασμολογικές προτιμήσεις, χώρες ΕΖΕΣ ή αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ε, ειδική προστασία από πλευράς Ένωσης. Τέλος, όπως σας είπα, πώς συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Αλληλεία. Έχουμε στην Γενική μας Διεύθυνση μια ομάδα που ασχολείται ακριβώ με τα θέματα αλληλεία. Είναι ειδικοί στον τομέα, ε, έχουν εμπειρία, είχαν δουλέψει στο παρελθόν και στη Γενική Διεύθυνση Αλληλεία. Η συνεργασία με την Γενική αυτή Διεύθυνση ήταν μέχρι τώρα πάρα πολύ θετική για μα. Μετέχει στη διαπραγματεύση η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και έχουμε δεσμ δεσμευόμαστε να συζητούμε μεταξύ μας πριν την αποδοχή της τελικής λύσης με τη, τελική τελικής ε, συμφωνίας με την τρίτη χώρα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον κλάδο, είμαστε σε μόνιμη επαφή με τον κλάδο για να ξεκινήσουμε, όταν ξεκινούμε νέες διαπραγματεύσεις θέτουμε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια στον κλάδο, ζητούμε από τον κλάδο να μας πει τι θέλει, ποια είναι τα συμφέροντα που θέλουν να ληφθούν υπόψη στο γύρο διαπραγματεύσεων, ενώ ταυτόχρονα μετέχουμε τακτικά στην Συμβουλευτική Επιτροπή Αλίας και Ιδετοκαλλιέργειας της Κομισιόν, όπου μας παρουσιάζει τις απόψεις του ο κλάδος, που λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων, όπως γνωρίζετε, πριν το ξεκίνημα οποιασδήποτε εμπορική ε, διαπραγμάτευση σε όλου του τομεί, όχι μόνο στην Αλία, γίνεται μια μελέτη αντικτύπου των διαπραγματεύσεων. Εάν η Ελία είναι σημαντικό κλάδο, όπω είναι για παράδειγμα στι διαπραγματεύσει με τι χώρε ΕΣΕΑΝ, είχαμε ειδική ανάλυση του αντικτύπου στον τομέα τη Ελία. Έτσι έχουμε μια πλήρη εικόνα των συνεπειών πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Αυτό ήθελα να σα πω. Ευχαριστώ. Δεν θα σας απαντήσω τώρα γιατί θα δώσω το λόγο στη στον κύριο Μπέιτς από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι στη, ο Ρίτσαρντ Μπέιτς ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και ζητώ συγγνώμη που ο κύριος Ραμόν δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Να σας πω πάντως ότι εδώ ακούστηκαν ορισμένα σημαντικά στοιχεία μέσα από τις τρεις πρώτες ομιλίες αλλά και μέσα από τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια οικονομική κρίση στην Ευρώπη και οι καταναλωτές ε, ξοδεύουν λιγότερα. Ταυτόχρονα, αυτό δεν είχε προβλεφθεί, δηλαδή ότι μια χώρα στην Ασία μέσα σε 7 χρόνια θα δημιουργούσε ένα νέο είδος που ε, πραγματικά ε, θα δημιουργούσε προβλήματα και σε σχέση και με την ηχθειοκαλλιέργεια ε, του, του σολομού, αν θέλετε, την εκτροφή σολομού. Έχουμε δηλαδή τώρα νέε παραγωγέ νέων προϊόντων που έρχονται στην αγορά. Ταυτόχρονα όμω είναι γνωστό σε και τον κόσμο ότι ε, εδώ από άποψη υγειονομική ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, και είχαμε και μια συγκεκριμένη ερώτηση του κ. Βαλέσα που μιλούσε για τα προϊόντα που έρχονται από την Κίνα και κατά πόσο ανηφίσατε του ίδιου ελέγχου με τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κοιτάξτε, από θα θυμάστε ότι από το 2002 στο 2004 δεν επιτρέπαμε τις εισαγωγέ προϊόντων αλίας από την Κίνα λόγω υγειονομικών προβλημάτων. Και μόλις το τέλος του 2004 άρχισαν, ε, άρχισαν πάλι να γίνονται εισαγωγέ. Πρώτα απ' όλα νοπών και, και πολύ αργότερα προϊόντα ηχθειοκαλλιέργειας. Άρα δεν είναι εδώ γίνονται έλεγχοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για διαφορές ε, σε οικονομικό επίπεδο και διαφορετική μεταχείριση. Όσον αφορά το άλλο στοιχείο που αναφέρθηκε για την βιωσιμότητα σε σχέση με το περιβάλλον και τα οικονομικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τα πρότυπά μας στους τομείς αυτούς, ε, με βάση, γιατί με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ δεν μπορούμε να πούμε στους παραγωγούς της Ασίας ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με την οδηγία Natura 2000, ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με την νομοθεσία που αφορά τα ύδατα, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Άρα εδώ βεβαίως υπάρχει διαφορά. Και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Άρα, τι κάνουμε. Πολλοί ομιλητέ είπαν, μίλησαν για την καθυστέρηση αυτή στη μεταρρύθμιση τη κοινή οργάνωση αγορά και ότι είναι απαράδεκτη. Ναι, θεωρήσαμε ότι ε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνδέσεις ε, ε της πολιτική ε, ε, πολιτικής με την αγορά, το καλύτερο που θέλαμε να κάνουμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε μια ολιστική προσέγγιση και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σε περισσότερο βάθο την κατάσταση. Για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα, την προσεχή εβδομάδα θα γίνουν δύο ξεχωριστά σεμινάρια για την πρόθεση και την προσφορά των ελληνικών προϊόντων ε, και προβλέπεται και ένα τρίτο σεμινάριο για τις ποιοτικέ πλευρές. Έχουμε αναθέσει επίσης μια νέα μελέτη των διαφόρων σεναρίων για την κατάσταση μέχρι σήμερα και το πώς η μεταρρύθμιση της οργάνωσης αγοράς μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανία. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η οργάνωση της ε, αγοράς πρέπει να ενισχύσει τους παραγωγούς, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των πόρων, ε, επικέντρωση της προσοχής στην, ε, στα ποιοτικά προϊόντα, καλύτερη σύνδεση των ε, προϊόντων με την αγορά, καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση και η ανάγκη οι καταναλωτές να έχουν τις σωστές πληροφορίες για τα προϊόντα λίας και, και ηχθειοκαλλιέργειας. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο θεμέλιος λήθος της μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι ε, περισσότερη ενδυνάμωση των οργανώσεων των παραγωγών, ε, ε, προσφορά και τι γίνεται με τις εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Και πώς τελικά ε, μπορούν οι καταναλωτές να έχουν τις πληροφορίες για τα προϊόντα μέσα από την σήμανση και την ανιχνευσιμότητα, γιατί αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε και το εξής γεγονός που έχει να κάνει με τις επιστημονικές πληροφορίες που καταδεικνύουν όλο και περισσότερο τα ωφέλη από την κατανάλωση ε, των προϊόντων της αλίας. Και στο μέλλον νομίζω ότι αυτό το, ε, ότι αυτό το προϊόν θα γίνει ε, λειτουργικό τρόφιμο, αν θέλετε. Δηλαδή, θα καταναλώνουν, ε, θα καταναλώνουν ψάρια για, για την, την υγεία τους. και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα ωμέγα λιπαρά, τα οποία περιέχονται περισσότερο στα ψάρια ανοιχτή θάλασσα και όχι στα προϊόντα ηχθειοκαλλιέργειας. εδώ, όσον αφορά τι ε, εμπορικέ διαπραγματεύσει για τα αλλιευτικά προϊόντα, η Γενική Διεύθυνση Εμπόριο έχει την ε, βασική αρμοδιότητα και όχι η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ, θάλασσα. Και να σα πω και το εξή. Ε, πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των μεταποιητών. Και τώρα θα έχουμε δύο μιλητέ από, από τον κλάδο τη μεταποίηση για να ακούσουμε και τους δύο κλάδους του, του τομέα. Και θα είναι σημαντικό να τοποθετηθούμε, αν μας δώσει την ευκαιρία πρόεδρε, και μετά από το δεύτερο αυτό πάνελ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να δώσω τώρα το λόγο στους τρεις ομιλητές. Σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, γιατί δεν πρόκειται να προλάβουμε. Αν θέλετε τώρα να κάνετε κάποια απάντηση, ο κύριος Τεϊχέρα έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τέθησαν πολλά ερωτήματα από όλους τους ε, ομιλητέ, και εγώ θα ήθελα ε, να ακούσω την άποψη τη ε, μεταποιητική βιομηχανία πριν τοποθετηθώ. Πάντω δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα. Ε, λοιπόν, και νομίζω ότι για παράδειγμα όσον αφορά την ε, ηχθειοκαλλιέργεια, ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βεβαίω ε, και πρέπει να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πρέπει να βελτιωθεί. Να αντιληφθούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Ότι τα ψάρια τρώνε ψάρια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ε, στις ζωοτροφές είναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Επίσης, εκτός από το καθεστώς των τιμών και τις εισαγωγές, και την κοινή οργάνωση αγοράς, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων των παραγωγών. Και να μην έχουμε αυτή την άκαμπτη στάση απέναντι στην εξέλιξη των αγορών. Να καταλάβουμε ότι οι εισαγωγέ δεν ε, αφορούν μόνο τι τιμέ αναφορά, αλλά και τα σχέδια διαχείριση των ίδιων των παραγωγών προσπαθούμε να διαχειριστούμε συγκεκριμένε ποσότητε και προσπαθούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις ποσοστώσεις σε κοινοτικό επίπεδο που θέλουμε να διαρκούν σε ολόκληρο τον χρόνο. Ε, για να μην έχουμε πρόβλημα τις αγορές και χρονικής διάρκειας. Αλλά ε, αυτό που έχετε σε αντίφαση με αυτή την ιδέα είναι αυτή η εισαγωγή προϊόντων Ε, που καταλαβαίνετε ότι ε, έχει να κάνει και με τις τιμές και με, και με τις ποσότητες. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με την οποία η αλία και με τους περιορισμούς που έχουμε σε επίπεδο τάκ και ποσοστώσεων. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις αγωγές, χρειαζόμαστε τις αγωγές, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να είναι συμβατά και με την ικανότητα ρύθμισης των δικών μας των αγορών στις δικές μας ζώνες αλίας. Ευχαριστώ. Κύριο Στίβενσον τώρα. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα στοιχεία που ακούσαμε σε ό,τι αφορά την ε, απόσυρση των σκαφών και του μακαλιάρου γαρίδας ε, στην ε, Σουηδία οφείλεται στα πολύ χαμηλότερα τάκ που ισχύουν και επίσης ε, στα μέτρα που λαμβάνουμε για την καλύτερη διαχείριση της αγοράς. Έχουμε και την πιστοποίηση μεσή. Όλα αυτά αποτελούν μέτρα που βελτιώνουν τη διάθεση στην αγορά. Όπως είπατε όμως, βρισκόμαστε αντίθετοι στο ρεύμα γιατί έχουμε τις ε, εισαγωγές τις ανταγωνιστικές και έτσι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το κέρδος παρά τις μειώσεις, παρά την πιστοποίηση της αλληλείας μας. Ουσιαστικά διατηρούμε το ίδιο επίπεδο τιμών με υψηλότερο κόστος, άρα χάνουμε περιθώριο κέρδους. Αυτό έχει να κάνει και με τους χαμηλούς ε, μισθούς που επικρατούν στον κλάδο. που επιτρέπουν στις περιοχές στους παραγωγούς να ε, έχουν πιο πολύ κέρδος ε, με τις τιμές. Είπατε ότι το μέλλον, στο μέλλον και για την επιτυχία της ΚΟΑ σημαντικό είναι το θέμα της πιστοποίησης και της επισήμανσης. Δεν Τέλος, ο κύριος Πισόν. Euh, euh, και εγώ θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία σε αυτό που ρώτησε η κυρία Λόβιν για τις αποσύρσεις. Κατά την άποψή μου, παρόλο που το πρόβλημα των αποσύρσεων είναι πρόβλημα το οποίο μας αφορά πρώτα απ' όλα εμάς. Γιατί αμφισβητώ ε, απόλυτα την ιδέα ότι οι ψαράδες πάνε να ψαρέψουν και το αντικείμενο της εργασίας τους να το πετάξουν στα σκουπίδια. Αυτό δεν ευχαριστεί κανέναν. Κυρίως αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν προφανώς πρέπει να βρούμε και άλλες λύσεις. Πιο ικανοποιητικέ. Η απόσυρση είναι το σύμπτωμα ε, του κακού και όχι το ίδιο το κακό. Το σύμπτωμα λοιπόν μιας ασθένεια που οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι κοινοτικοί αλληλείς δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη μείωση των τιμών που νομίζω ότι σας την έδειξε και πριν από λίγο γιατί πλέον δεν θα είναι αποδοτική για αυτούς η εργασία τους. Το σύστημα λοιπόν που εφαρμόζουμε οδηγεί σε μια κατάσταση όπου θέτουμε ελάχιστες τιμές ε, πέρα των οποίων αρνούμεθα να απολύσουμε το προϊόν διότι δεν είναι πλέον αποδοτικό. Αλλά βλέπουμε και εδώ υπάρχουν και άλλες αιτίε και εδώ σας παραπέμπω και στην παρέμβαση της εκπρόσωπου της Γενικής Διευθύνση Εμπορίου. Αυτή ε, η διαφορά ανταγωνισμού είναι τόσο μεγάλη που Βεβαίω, αν καθορίσουμε τη μέσα σε, ε, σε υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια τιμή, δεν θα μα οδηγήσει αυτό πουθενά. Αλλά όταν, μας, όταν ακούμε ότι οι εισαγωγέ είναι απαραίτητε, βεβαίω δεν πρόκειται προ Θεού ε, να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά όταν ακούμε ότι μια μελέτη που τη γνωρίζω άλλωστε του Μαΐου του 2009 δείχνει ότι αυτό δεν έχει επίπτωση στην κοινοτική παραγωγή, τώρα μα λέτε ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ έχουμε παρεστήσει και ότι οι μειωμένε τιμέ που ζούμε δεν υπάρχουν. Ε, μα δυστυχώ υπάρχουν. Αν θέλουμε να καταστήσουμε ε, τους κοινοτικούς τόλους πιο ανταγωνιστικούς, και σας το έδειξα πριν από λίγο, το κόστος εργασίας ε, στα ε, ε, κοινοτικά πλοία ε, διαφέρει σημαντικά από το κόστος ε, των τρίτων χωρών που είναι στο 30-35% του κοινοτικού. Άρα λοιπόν, πρέπει, αν δεν θέλουμε να μειωθούν οι τιμές, πρέπει να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών. Το να λέτε λοιπόν σήμερα ότι θα μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί, δεν να μην σας πω ότι είναι προσβολή, αλλά Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικά καθόλου αυτά, άρα κατά κάποιο τρόπο μας, αυτά είναι κοροϊδίες. Και τελειώνω. Με την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Θάλασσα. Σε αυτή την ιδέα δηλαδή ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε περιβαλλοντικούς ε, κανόνες ε, στους υπόλοιπους. Βεβαίως, οι ε, κοινοτικέ οδηγίε εφαρμόζονται στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Natura 2000 δεν μπορεί να το εφαρμόσει το Βιετνάμ. Φυσικά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για κοινοτικά πρότυπα. Μιλάμε για δεσμεύσει που ελήφθηκαν ε, με συνένεση όλων των συμβαλωμένων μερών του ΟΗΕ. Η σύσταση 30 ε, τη Συνόδου Κορυφή του Johannesburg, που μα λέει ότι το 2015 το πολύ τα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο διαχείριση σύμφωνα με τι μέγιστε βιώσιμε αποδόσει. Βεβαίω θα μα πείτε ότι και εμεί εδώ στην Ευρώπη, όσον αφορά ορισμένα αποθέματα, δεν έχουμε πετύχει το στόχο αυτό, αλλά έχουμε τα μέσα και όταν μιλάω για ληφτικά πρότυπα, εδώ αναφέρομαι. Ποια είναι τα μέσα ε, αξιολόγησης ε, των αποθεμάτων, άρα διάγνωσης, και δεύτερον ε, εφαρμογή μέσων διαχείρισης. Στην Ευρώπη, όταν η κατάσταση ε, ενός αποθέματος, των αποθεμάτων ενός είδους δεν είναι γνωστή, εφαρμόζουμε μία κλίμακα που περιέχεται στο έγγραφο ε, πολιτικού προσανατολισμού και που καθορίζει το είδο των κανόνων που θα εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο απόθεμα, στο μέτρο που η κατάσταση είναι άγνωστη. Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να αυξήσουμε ε, την αλληλευτική ικανότητα. Υπάρχει αυτό το policy statement, το οποίο κάθε χρόνο καθορίζει του κανόνε που εφαρμόζονται σε διάφορα αποθέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναρτήσει τη κατάσταση. Είτε πρόκειται για ε, επιδείνωση του αποθέματος είτε όχι. Αυτό υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλοι αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση. Αν οι ποσοστώσει μα μειώνονται κάθε χρόνο, αν οι ελευτικέ ικανότητε μειώνονται κάθε χρόνο, αυτό οφείλεται σε αυτού του κανόνε. Τι εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση απλά και μόνο να επαληθεύσει ότι στι χώρε που εξάγουν προϊόντα αλληλευτικά ε, θα υπάρξουν ανάλογοι κανόνες. Δεν λέμε ότι θα ακολουθήσουμε τους ίδιους κανόνες διαχείρισης και εκεί, αλλά ότι θα έχουμε κάποιες βάσεις. και θα έχουμε εξασφαλίσει ότι οι βασικοί αυτοί κανόνες αφορούν και αυτά τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μία απάντηση σε μια ερώτηση που έγινε σχετικά με τα λεφτικά πρότυπα. Ευχαριστώ. Κατ' εξαίρεση, καθότι ήταν εισηγητή, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρέκο που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτό το εξαιρετικό μέτρο που λάβατε. Ήθελα απλά να πω ότι όσο περισσότερο σας ακούω συνάδελφοι, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι η έκθεση που μου αναθέσατε είναι αναγκαία. Πολλά από τα ερωτήματα προς την Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνουν αυτά που υπήρχαν στο κείμενο εργασία που σας υπέβαλα πρόσφατα. Αντίθετα, ωστόσο, οι απαντήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου δεν με έπεισαν. Θα επανέλθω και θα επαναλάβω αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Πίσω. Λέτε ότι οι εισαγωγέ δεν έχουν αντίκτυπο στις τιμές. Ίσως για κάποια είδη το λαβράκι. Αλλά για πολλά άλλα αυτό δεν ισχύει ουδόλως. Είναι πασιφανές αυτό. Ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές, του κύριο Τεσέιρα Πίσον και Στίβεσον για τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Οι τελευταίοι ομιλητές, δύο εκπρόσωποι του κλάδου του, της διανομής. Ποιος από τους τρεις είναι έτοιμος να μιλήσει δεν ξέρω. Ο κύριος Κέλλερ, ο δόκτωρ Κέλλερ, εκπρόσωπος της, ενώσης, ε, της Ενώσεως μεταποίηση της και του Εμπορίου ε, σε χονδρική του χονδρεμπορίου στην αλεκτικό πρόεδρο στη Γερμανία. Τον ξέρουμε, έρχεται συχνά, τον ευχαριστούμε γιατί είναι τακτικός θαμώνας της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο κύριε Κέλλερ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισηγητή, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ πέρα ως εκπροσώπους της ε, μεταπητικής βιομηχανίας. Θα ήθελα να σας καλέσω στην παρουσίασή μου να, κάνουμε μια, να κοιτάξουμε τι γίνεται σε 6 χρόνια, στο 2015. Θα ήθελα να σας πω ότι 16 εκατομμύρια τόνοι θεωρώ ότι θα είναι η προσφορά ψαριού στην Ευρώπη και 4 εκατομμύρια θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία για την Βιτοκαλλιέργεια, 1,5 εκατομμύριο και 10 εκατομμύρια τόνοι από εισαγωγέ για να ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση. Δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε στο μέλλον χωρί τι εισαγωγέ ή θα πρέπει να μειώσουμε την ε, κατανάλωση. Αυτό τι σημαίνει, ότι στο τραπέζι μα, στο πιάτο μα το 2015 θα έχουμε κατά ένα τέταρτο προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Αλληλεία, 10% από την καλλιέργεια και κυρίε και κύριοι 76-75% πάνω από 2 τρίτα θα προέρχονται από εισαγωγές. Δεν μπορώ να σας διευκρινίσω πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τότε, αν θα πρόκειται για ψάρια από υδατοκαλλιέργεια ή όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα αυξηθεί το ποσοστό της υδατοκαλλιέργειας. Δεν χρειάζεται να σας πω γιατί θα διευρυνθεί η αγορά. Έγραψα κάποιους από τους λόγους που πιστεύω ότι θα ισχύουν, αλλά νομίζω ότι και εσείς, ε, ίσως όχι κάθε μέρα, αλλά πλέον δύο φορές την εβδομάδα, τρώτε ψάρι. Είτε εδώ, είτε στην ε, εκλογική σας περιφέρεια και ξέρετε τι λένε γιατροί, ότι χρειάζεται και το λιπαρό ψάρι και το πιο λιγότερο λιπαρό ψάρι και ξέρετε εσείς κυρίες μου ότι το ωμέγα 3 είναι καλύτερο από κάθε αντιγυραντική κρέμα και για τους άντρες ασφαλώς ε, είναι καλό το ωμέγα 3, όχι μόνο για τις γυναίκες. Και να θυμάστε πάντα στα πάρτι να τρώτε και λίγο σε Σκουμπρί. Σκουμπρί. Θαύματα κάνουν αυτά τα ψάρια. Τώρα, για αυτό το ισότιμο επίπεδο, το 11 playing field, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία από πλευράς ε, των αλλιέων και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση για το μέλλον. Δεν είναι εξαιρετική. Να σας τα παρουσιάσω όμως τα στοιχεία αυτά για να μην τα ξεχνάτε στις μελλοντικές σας συζητήσεις. Καταρχάς, το MSY. Ε, πολύ σωστό για την βιώσιμη αλληλεία μέχρι το 2015 θα έχει συνέπειες για τα πιο πολλά είδη σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις που ορίζονται στην Ευρώπη. Είναι σαφές κυρίες και κύριοι ότι το ψάρι πάντα νοπό το ψαρεύουμε. Και το ψαρεύουμε και ολόκληρο. Δεν το ψαρεύουμε σε φιλέτα. Αλλά τι ζητάει η αγορά και τι θα ζητάει η αγορά στο μέλλον. Στο μέλλον, ξέρετε, θα επικρατήσουν τα πιο άνετα συσσαγωγικά προϊόντα, τα φιλέτα. Τα φιλέτα αυτά πώς προκύπτουν με την πρώτη μεταποιητική φάση. Εκεί διαπιστώνουμε ότι η πρώτη αυτή μεταποίηση και αυτή δεν λαμβάνει πλέον χώρα στο ιστορικό το, της Ένωσης, γιατί δεν έχουμε εργατικό δυναμικό που ξυπνάνε πρωί-πρωί μέσα στα, στη μαύρη νύχτα για να ετοιμάσουν τα φιλέτα αυτά. Άρα και αυτή η πρώτη μεταποίηση έχει μετακατασταθεί εκεί που υπάρχει το εργατικό δυναμικό και ο συνάδελφος Πισό μας εξήγησε τι σημαίνει αυτό για το κόστος. Αλλά, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε να μην πέφτετε στην παγίδα τέτοιων εύκολων υπολογισμών και μόνο η παρουσίαση του απόλυτου κόστους δεν σημαίνει ότι μια βιομηχανία, ένας κλάδος είναι ανταγωνιστικός. Θα πρέπει να κοιτάξετε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ω προς το κόστος και στο πλαίσιο αυτό να δούμε και την παραγωγικότητα, την εργατική παραγωγικότητα. Αν δεν λάβουμε υπόψη τις ε, συνιστώσεις αυτές, δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε τους μισθούς. Ε, τα 20 δολάρια ανά ώρα, 108 δολάρια, δεν ξέρω αν ημέρα κτλ. Είναι πολύ απλοϊκές αυτές οι συγκρίσεις. Επίσης θα υπάρχει έντονη τμηματοποίηση των αγορών. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πώς θα καταναμηθεί η κατανάλωση νόπου και κατεψυγμένου ψαριού. Και τα τελευταία δύο στοιχεία τώρα. Θα υπάρξει περιορισμός ε, της παραγωγικότητας και της δυνατότητας προμήθειας της Ευρωπαϊκής Αλληλείας, γιατί καταρχάς έχουμε τις ζώνες των 200 μιλίων που έχουν εισηχθεί πριν από πολλά χρόνια και κατά δεύτερον υπάρχει και ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις, ε, τους πόρους. Να περάσουμε εν συντομία στα θέματα της υδατοκαλλιέργειας, τα οποία έθιξε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Και εδώ είναι σαφές ότι δεν θα μετρήσει μόνο το απόλυτο κόστος, αλλά και το συγκριτικό κόστος και το συγκριτικό κόστος θα είναι υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν η υδατοκαλλιέργεια δεν πρόκειται να ωφεληθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Κατά δεύτερον στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες γεωγραφικά ευνοημένες περιοχές για υδατοκαλλιέργειες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο ευνοημένες όσο ε, περιοχές, χώρες του νοτίου ημισφαιρίου. Και όλοι γνωρίζετε τι γίνεται με τους κύκλους παραγωγής. Αν ε, είναι καλές οι τιμές, υπάρχει μεγάλη παραγωγή και το βλέπουμε αυτό να ισχύει και με τους χείρους, για παράδειγμα. Όταν πέφτουν οι τιμές, μειώνεται και η παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τα ψάρια. αυτό για μια μεταποιητική βιομηχανία η οποία χρειάζεται μια σταθερή ροή είναι απόλυτα ε, αποσταθεροποιητικό. Και αυτό θα επιβαρύνει την ευρωπαϊκή ηθοδοκαλλιέργεια και κυρίες και κύριοι αν προσπαθήσουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταστήσουμε μια τέτοια υδατοκαλλιεργική μονάδα θα διαπιστώσουμε ότι είναι τόσο υψηλά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που θα σταματήσουμε την προσπάθεια μετά από λίγες εβδομάδε. Να κοιτάξουμε την μεταπητική βιομηχανία τώρα. Στην παρούσα φάση μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η ζήτηση που έχουμε ικανοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει και να εξακολουθήσει να ισχύει και στο μέλλον. Ό,τι αγοράζουμε λοιπόν από τρίτες χώρους, χώρες, συγγνώμη, δεν ε, αγοράζονται δίχως προδιαγραφές. Όχι. Αγοράζονται μόνο τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα. Με προσανατολισμό πάντα στη ζήτηση. Και τα παραδοσιακά είδη ψαριών, τα οποία είναι ανταγωνιστικά, αν θέλετε, αντιμετωπίζουν το πλανέκτημα στις εισαγωγές γιατί με τις εισαγωγές αν θέλετε μπορούμε να εισάγουμε πολλά και διαφορετικά ψάρια. Μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονό ότι αναφέρετε ότι θέλετε κι εσεί να τα ρυθμίσετε αυτά. Κοιτάξτε το 4. Οι καταναλωτέ απαιτούν από εμά σήμερα νέα προϊόντα. Τα νέα προϊόντα, αυτά μπορεί να είναι προϊόντα, ξέρετε, ε, άνετα εισαγωγικά που εξοικονομούν χρόνο, αλλά και απλά προϊόντα τα οποία δίνουν μία εγγύηση. Τι εγγύηση εννοώ. Μία εγγύηση, για παράδειγμα, με την σήμανση MSC η ζήτηση για προϊόντα MSC δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από ευρωπαϊκές πηγές. Χρειαζόμαστε εισαγωγές προκειμένου να εισάγουμε τέτοια βιώσιμα προϊόντα. Και να σας πω ότι στο μέλλον θα έχουμε και το, τη σήμανση ASC για τις υδατοκαλλιέργειες η οποία θα επικρατήσει. Να δεν μπορώ παρά να παροτρύνω τους ε, υδατοκαλλιεργητές ε, στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για τα πρότυπα αυτά για είδη όπως ο Παγκάσιος και ο Τιλάπια. Ακούσαμε πολλές φορές ε, και είπε και ο συνάδελφος Στίβενσον ότι εισάγονται χαμηλής ποιότητας ψάρια. Κυρίες και κύριοι, πιστεύετε πραγματικά ότι εκατομμύρια α, ε, αγοράζουν παγκάσιο κάθε μέρα κατά λάθο επειδή είναι κακής ποιότητας. Καλά, άμα το πιστεύετε, έχετε ίσως μια καλή αντίληψη για τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι Πρόκειται για μια καλή λύση, για ένα γεύμα, για μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτή. Μιλάμε για την ελάχιστη τιμή. Αλλά να σας υποδείξω ότι υπάρχει και μια άλλη τιμή. Κοιτάξτε την τιμή για λευκά προϊόντα με φτερούγες ως επιτεπλίστων. Για το κοτόπουλο. Τα πουλερικά. Αυτό αποτελεί την τιμή ορόσημο για τα προϊόντα μας. Όχι η τιμή για την πεσκανδρίτσα και το λαβράκι. Και είμαι πεπισμένος κυρίες και κύριοι ότι μακροπρόθεσμα οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μας πάρουν τα ψάρια και θα αυξηθούν οι τιμές του ψαριού. και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει μια ευκαιρία για τους ε, Ευρωπαίους αλληλείς. Κοιτώντα την μεταρρύθμιση τη κοινή ελεκτική πολιτική, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη τα εξή στοιχεία. Καταρχά, ότι χρειαζόμαστε ένα φιλελεύθερο ε, καθεστώ εισαγωγών για τις πρώτες ύλε, Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε στον ανταγωνισμό να επιβιώσουμε με ευρωπαϊκό προϊόντα, γιατί θα έχουμε προβλήματα και με τα επιδοτούμενα προϊόντα, όπως το κοτόπουλο. Επίσης, λέτε, κύριε Σιγητά, ότι θέλετε να μετατεθούν οι αρμοδιότητες στην Γενική Διεύθυνση της Θάλασσας. Εμεί κοιτάξτε, όχι δεν συμφωνούμε. Εμεί προτιμούμε τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου γιατί διαβουλεύεται μαζί μα μας αφήνει να συμμετέχουμε στι εξελίξει, Είναι εξαιρετική η συνεργασία και την επιθυμούμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι αυτονόητο κυρίε και κύριοι ότι οι κανόνε προέλευση θα πρέπει να τηρούνται σε όλε τι εισαγωγέ και ακούσαμε ότι γίνονται εισαγωγές χαμηλή ποιότητα ψαριού, κύριε και κύριοι. Υπάρχει ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τις εισαγωγές. Κάθε εισαγωγή ελέγχεται με συστηματικό τρόπο. Να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτό πού σημαίνει στις ε, φορτώσεις. Είναι όλα τα ψάρια δηλαδή των Ευρωπαίων παραγωγών ε, ε, ελεύθερα από δύο ξύνες, από ισταμινικά κτλ. Είναι όλα δηλαδή εγγυημένης ποιότητας. Ζητώ λοιπόν ένα σύστημα γρήγορη πρατοποίηση και τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και επίσης ξέρουμε κάθε μήνα τι εισαγωγέ έγιναν. Οι μηνιαίες όμως στατιστικές για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που είναι. Δεν υπάρχουν. Και βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει διαφορά και ότι υπάρχει μειονέκτημα. Δεν εισάγουμε όμως ε, ψάρια και δεν υπάρχουν σχετικέ ε, επιδοτήσει, το οποίο μου φαίνεται ε, λογικό. Σας ζητώ εδώ πέρα στην Επιτροπή Αλληλεία να υπάρξει μια πιο ε, συνεπής ορολογία σε ό,τι αφορά τις νομικές προδιαγραφές, γιατί είναι πραγματικά εφιαλτική η κατάσταση. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα που θα πρέπει πραγματικά να πάρει ένα τέλο αυτή η κατάσταση. Δεν χρειαζόμαστε πιο πολύ ρύθμιση, χρειαζόμαστε λιγότερη ρύθμιση και ο κανονισμό για την επισήμανση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω και να ρωτιέμαι σε πόσα κράτη έχει εφαρμοστεί πλήρω. Σα παρακαλώ λοιπόν να μην δημιουργούμε διαρκώ νέα νομοθετήματα, αλλά να ελέγχουμε την εφαρμογή των παλιών. Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω και το εξή ότι και στο μέλλον θα χρειαστούμε την υποστήριξη για το promotion, για την διάθεση στην αγορά. Και καλό θα ήταν στο σημείο αυτό να μην υποχρεώνονται μόνο για συγχρηματοδότηση τα κράτη-μέλη, αλλά να έχουν μια ανώτερη εποπτεία σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση και να μπορεί να μπορούν τα χρήματα αυτά να προέρχονται και από τους εμπλεκόμενους φορείς, όταν πρόκειται για τέτοιο γενικό μάρκετινγκ. Τέλος, να μην ξεχνάμε το θεώρημα του Ντάβιτ Ρικάρντο, ο οποίος είχε πει κάποτε ότι το συγκριτικό κόστος και έχουμε και ένα σχετικό έγγραφο της ΦΑΟ πλέον, το οποίο σας συστήνω να διαβάσετε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μίλησα λίγο παραπάνω από το χρόνο που μου έχετε δώσει, αλλά προσπάθησα να τηρήσω τελικά το χρονικό περιθώριο. Ευχαριστώ κύριε Γκέντερ. Ε, πραγματικά ήσασταν προκλητικός με τις ερωτήσεις σας ε, και με τις ερωτήσεις που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαξουίν, εκπρόσωπο της ε, Ομοσποδίας ε, Αλλιέων της ε, Σκοτίας. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Good morning, Chairman. Thank you very much. It's always a bit of a... Ευχαριστώ. Πάντα είναι πρόβλημα. όταν εφόσον μίλησε πρώτα ο κύριος Σκέλλερ Χαίρομαι όμως γιατί ε, μίλησε ε, για το ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, κατανάλωση αυτών των, των ψαριών, το σκουμπρί και της ρέγκας. Κοιτάξτε, εδώ κατά κάποιο τρόπο έχω, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Οργάνωση των παραγωγών, αλλά θα έπρεπε να είχαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ντόναχιου. Έχω πάρει τη θέση του, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν, να σας ε, μιλήσω για την ευρωπαϊκή οργάνωσή μας. Εκπροσωπούμε οργανώσεις παραγωγών από 10 κράτη-μέλη. 10.000 περίπου είναι τα σκάφη μας, από μικρά μέχρι ε, μεγάλες ε, τράτες καταψύκτες. Ετήσια η συνδυασμένη παραγωγή αυτών των πλοίων είναι 3,5 εκατομμύρια τόνους ενώ οι πωλήσει ανέρχονται ε, σε αξία 3 δις ευρώ το χρόνο. Μας ε, απασχολεί ιδιαίτερα η κοινή οργάνωση της αγοράς και το πώς θα εφαρμοστεί. Και ο κύριος Κέλλερ μας ε, έδωσε μία εικόνα και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Εγώ θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα και να σας μιλήσω για τα, για τα προηγούμενα δέκα χρόνια και τι μας έφεραν. Ο κανονισμός 104-2000 είναι το νομικό μέσο που επιτρέπει την ίδια την δημιουργία των, των οργανώσεων της αγοράς. Η μεταρρύθμιση του λοιπόν είναι κρίσιμη σημασίας για την ίδια μας την ύπαρξη και για το ρόλο που θα παίξουμε. Και όπως αναφέρει και ο κανονισμός, οι οργανώσεις των παραγωγών αποτελούν το θεμέλιο λίθο, τη ρεχοκοκαλιά της κοινή οργάνωσης αγοράς. Αυτό αναγνωρίζει σαφώς την ανάγκη οργάνωση των παραγωγών, των αλλιέων, συγγνώμη, με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να ε, αντισταθμίζουν ε, τις, ε, του, τους μεγάλους μεταποιητές και τους ακόμη μεγαλύτερους λιανέμπορους. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός θεσπίζει ότι οι οργανώσεις των παραγωγών θα πρέπει να μπορούν να συγκεντρώνουν την προσφορά στην αγορά. Αυτό το οποίο όμως είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια κατά την άποψή μου είναι ε, να αποδίδεται ε, όλο και μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις ε, απαιτήσει. Αυτό το 2000 είναι ακόμα περισσότερο αλήθεια σήμερα. Ο κανονισμός του 2000 αναφέρεται στο γεγονός ότι οι αλληλείς αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση ε, προσφοράς. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε την τελευταία δεκαετία είναι ότι αυτή η συγκέντρωση ε, κλιμακώθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό. Και τώρα η κατάσταση είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι μία ε, από τις μεγαλύτερες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο στα διαταλλευτικά προϊόντα. 66,5 δις δολάρια το χρόνο έχει υπολογιστεί ότι αντιπροσωπεύει ε, η αγορά αυτή. Μεγαλύτερο λοιπόν από τα 65 ε, δις ε, δολάρια το χρόνο της Ιαπωνίας που ήταν μέχρι τώρα ο μεγαλύτερος καταναλωτής αλλιευτικών προϊόντων. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ σημαντικός παίκτη στην παγκόσμια αγορά αλίας. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αλλαγές, ραγδαίες αλλαγές, μαζικές αλλαγές που επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο αλλιεύουν ε, και μεταποιούν ε, τα προϊόντα οι αλλοίς. Η φρικτή λοιπόν παγκοσμιοποίηση έφτασε στην αλληλεία νωρίτερα από ό,τι σε άλλους τομείς. το προβλήματα όμως τα οποία συνδέονται με το φαινόμενο αυτό δεν μπορούν κατά την άποψή μας να επιληθούν με τον υφιστάμενο κανονισμό τα, ε, τα, οι παραδοσιακέ μέθοδοι αλληλεία και μεταποίηση έχουν αλλάξει και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ε, και έχουν αλλάξει ριζικά και αυτό έχει σοβαρέ επιπτώσεις για ολόκληρη τη βιομηχανία. Όπως ε, ε, είδαμε και τα τελευταία χρόνια με τη στασιμότητα των τιμών και με την αύξηση του κόστου λειτουργίας. Ελπίζουμε ε, αυτό, ε, ε, η μείωση των λευτικών αποθεμάτων να είναι προσωρινή. Αλλά αυτό οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των εισαγωμένων προϊόντων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι εξακολουθούν να γίνονται ορισμένες εξαγωγές. Μόνο που δεν συγκρίνονται με τις μαζικές εισαγωγές. Με μεγάλη μου λύπη λοιπόν παρατηρώ ότι η βασική παραγωγή της σκοτίας, ρέγκας δηλαδή και σκουμπριού, ε, σε μεγάλο βαθμό αποτελεί ε, αντικείμενο εξαγωγής. Άρα λοιπόν πρέπει να μας βοηθήσει και ο κύριος Κέλλερ για να ε, προσελκύσουμε τον Ευρωπαίο καταναλωτή να καταναλώνει περισσότερο σκουμπρί και περισσότερη ρέγγα και να μην κάνουμε αυτές τις εξαγωγές. Η άλλη βασική αλλαγή που έλαβε χώρα και που αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ είναι το γεγονός ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή βρέθηκε στο επίκεντρο ε, της μεταποίησης και αυτό έχει να κάνει ε, με, το, με τους νέους τρόπους αλίας. Και όπως είπε και εκπρόσωπος της Επιτροπής, χώρες όπως το Βιετνάμ, που δεν έκαναν καθόλου εξαγωγέ ε, αλληλευτικών προϊόντων ε, ε, πριν από λίγα χρόνια. Τώρα έχουν αυξήσει μαζικά τι εξαγωγέ, κυρίω του Παγκάσιου. Και από ό,τι κατάλαβα, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο Βιετνάμ απασχολούνται στον τομέα τη αλληλεία ενώ 5 ε, δις ε, δολάρια ε, το χρόνο είναι οι εξαγωγές. Και μία από τις βασικές αγορές εισαγωγής αυτών των προϊόντων από το Βιετνάμ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτές τις δραματικές αλλαγές στην αλληλεία στην, και στη μεταποίηση, το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή οργάνωση της αγοράς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Η αλληλείς από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν και όπου μπορούσαν να έχουν μια κάποια επίδραση στις τιμές, βρέθηκαν σε μια κατάσταση όπου πραγματικά ε, ακολουθούν την κατάσταση με παθητικό τρόπο. Έχει υπάρξει μεγάλη μετατόπιση υπέρ της μεταποίησης και της κατανάλωσης. Ε, για να σας δώσω μια ε, εικόνα. Το 2010 η αύξηση ε, στην, ε, στη θάλασσα του Μπάρεντς κατά 49.000 49 ε, τόνους είναι μεγαλύτερη από την αλία του, του γάδου στην, συνολικά στη Βόρεια Θάλασσα. Δηλαδή μιλάμε για συγκέντρωση σε ένα πολύ μικρό σημείο. Ο, ο κανονισμός του 2000 και η κοινή οργάνωση αγοράς έχει θέσει, ένα, ε, ε, ε, έχει θέσει ορισμένους στόχους. να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση, να σταθεροποιήσει τις τιμές και να εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος του Σαλή και να προωθήσει τη γενική ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου στι παγκόσμιες αγορέ. Δυστυχώ, ο κανονισμό δεν, δεν είναι επαρκή για την επίτευξη των στόχων αυτών, διότι αφορά μια διαφορετική περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν ε, ε, όλα αυτά τα θέματα ε, στο παρελθόν. Η συνολική διαδικασία καθορισμού τιμών αναφοράς πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά χρησιμοποιώντας πραγματικά και ρεαλιστικά στοιχεία. Η ελλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρόσφατα χρόνια. Και οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ε, παρέμβαση θα πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το φως της σημερινής κατάστασης στον τομέα προσφορά και ζήτησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει ε, κανείς αυτή την προώθηση ε, των ποιοτικών προϊόντων όταν από την άλλη υπάρχει πείνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, Βεβαίω ε, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και η οργάνωσή μα είναι έτοιμη να αρχίσει ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι τεχνικέ πτυχέ, παράδειγμα μεταφορά πρηματοδοτήσεων κτλ. Και το πώ αυτά μπορούμε να τα λύσουμε με καλύτερο τρόπο τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι ήδη ελέγχθη ότι ο κλάδος αλίας πρέπει να αναγνωρίσει ότι θα πρέπει να ε, γίνονται εισαγωγές για να αντιμετωπίσουμε το ε, ε, το θέμα της ζήτησης. Δεν ξέρω κατά πόσον οι προβλέψεις του δόκτωρα Κέλλερ θα εκπληρωθούν, γιατί κάτι το οποίο ανέφερε και το οποίο είναι σημαντικό και το ανέφερε στο τέλος της παρουσίασής του, είναι ότι οι αναδυόμενες χώρες αρχίζουν να αυξάνουν τη δική του ζήτηση για τα προϊόντα Και όσο θα αυξάνεται η ζήτηση αυτή, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ε, λιγότερες εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο και στις τιμές. Αλλά δεν θα πρέπει πάντως ε, αυτά τα προϊόντα εισαγωγής να είναι το απο, να οδηγούν ε, στο να διώξουν ε, τους ε, αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις, από τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να υπάρξει μια πιο σωστή ισορροπία. Και κοιτάξτε, όσοι ασχολούμαστε με την αλληλεία βλέπουμε κάπως ηρωνικό το θέμα ότι η Ισλανδία και η Νορβηγία που είναι οι βασικοί ε, ωφελούμενοι από την κοινή οργάνωση της αγοράς δεν είναι μέλος ε, της ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερα τις αλλαγές που έλαβαν χώρα ε, σε διεθνές επίπεδο ε, ε, όσον αφορά το πού γίνεται η αλεία, πού γίνεται η μεταποίηση και πού γίνεται η κατανάλωση. Ταυτόχρονα όμως έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της εταιρικής ευθυνη Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, κυρία Πρόεδρε, ότι η αηφορία και η ανιχνευσιμότητα είναι ε, τώρα ε, στο επίκεντρο, των, ε, στο επίκεντρο του καταναλωτή και των επιθυμιών του. Αλλά αυτοί οι στόχοι δεν αναφέρονται πουθενά στον υφιστάμενο κανονισμό της κοινή οργάνωσης αγοράς. Δεν αναφέρονται καν. Υπάρχει κενό δηλαδή το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της νομοθεσίας, διότι δεν αντιμετωπίζεται ένα θέμα το οποίο είναι τόσο μεγάλη σημασία. Form Αυτά τα σημεία πάντως σίγουρα θα πρέπει να αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης. Και είναι κάπως ηρωνικό το γεγονός ότι οι αλληλείς αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώνουν ε, για την εικόνα του προϊόντος τους πριν καν μπορέσουν να το πουλήσουν. Όταν μιλάμε για αποθέματα τα οποία ε, καλύπτουν την κοινή ελευτική πολιτική τουλάχιστον να ελπίσουμε ότι η μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς που ε, ε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ο κύριος Ογκάλαχερ το ανέφερε όχι σε τρία-τέσσερα χρόνια, ε, σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτική πολιτικής θα οδηγήσουν σε ε, αύξηση της εικόνας ε, του προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι προέρχεται δηλαδή από βιώσιμα αποθέματα και ότι τίθεται ανάλογα σε εμπορία. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα πρέπει να συμπεριλάβει κάποια μορφή οικολογικής σήμανσης, ε, γιατί αυτό ζητούν οι βασικοί αγοραστές και οι καταναλωτές. Ο καταναλωτής θέλει να αγοράζει προϊόντα οποία πληρούν τα πρότυπα αυτά. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα εν συντομία να σας πω ότι ενώ ε, από τη μια θα θέλαμε ένα ιδεώδη κόσμο με ένα ε, απόλυτα ελεύθερο σύστημα, ε, αυτό όμως ε, θα μπορούσε να οδηγήσει ε, σε πλήγμα κατά, της, κατά του, ιστορικού, κλάδου. Η ασφάλεια ε, στον προϊόντων διατροφής θα αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για όλες μας τα επόμενα χρόνια. Γίναμε, αν θέλετε, μια αστική κοινότητα. Έχουμε όμως πλούσιες, ε, πλούσιους πόρους ε, στις θάλασσες και στη γη μας. Αν καταστρέψουμε τη βιομηχανία που έχουμε σήμερα και που ε, μας βοηθά ε, να προβαίνουμε στην κομιδή αυτών των προϊόντων, τότε δεν θα μπορούμε πλέον να, να, δίνουμε αυτή την πρωτεΐνη υψηλή ποιότητα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κέλλερ και την οποία ζητούν απεγνωσμένα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μαξίν για την παρέμβασή σας και γιατί τηρήσατε και το χρόνο σας. Τελευταίος, ο κύριος Χουάν Μανουέλ Βιέιτης Μπαπτίστα Ντεσόσα, Γενικός Γραμματέας των Κονσερβοπαραγωγών της Ισπανίας. Έχετε το λόγο και εσείς για 15 λεπτά. Gracias, Presidenta. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Αιλίας του Κοινοβουλίου για την πρόσκληση που μου ευθύνεται και την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας. Να σας πω καταρχάς ότι η οργάνωσή μου, η Αμφάκο, είναι ε, μια, επιχειρη... μια οργάνωση επιχειρήσεων του 1904. Άρα έχουμε μια ζωή 106 ετών καλύπτει όλο τον κλάδο μεταποίησης ε, ε, από όλες τις ε, νοπά, κατεψυγμένα, όλα τα μεγάλα είδη βακαλιάρου, αλλά και της βιομηχανίας του τόνου. Και μάλιστα είμαι πρόεδρος και της Euratun που είναι η οργάνωση των σκαφών που αλλιεύουν τόνο στην Ευρώπη περιλαμβάνουμε γύρω στις 130 επιχειρήσεις με 4,5 δις κύκλο εργασιών. Θα σταθώ στα βασικά θέματα της ε, παρουσίασής μου, την κοινή αλληλευτική πολιτική και το εμπόδιο, το εμπόδιο συγγνώμη, και την αγορά. Να τονίσω ότι θα σταθώ στη σημασία πρώτα πρώτα της μεταποιητικής βιομηχανίας της Αλίας και της Ιδωτοκαλλιέργειας στην Ευρώπη των 27, τα χαρακτηριστικά για την Ισπανία και ιδίω για την Γαλλικία που είναι η πιο σημαντική περιοχή, τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης και τους στόχους της κοινή ελευτικής πολιτικής, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων συμπερασματικού χαρακτήρα. Να σας πω καταρχάς ότι η κοινοτική βιομηχανία σε επίπεδο του 27 με βάση τα στοιχεία της Eurostat και με άλλες πηγές. Έχει γύρω 4.000 επιχειρήσεις, 658 από αυτές στην Ισπανία, 204 από αυτές στην Γαλλικία. Άρα περίπου το ποσοστό της Ισπανίας στην Ένωση είναι 16%. Αφορά Υπάρχουν στην Ένωση 130.000 εργαζόμενοι στον κλάδο, 22.798 στην Ισπανία, ενώ στη Γαλλικία που είναι η κύρια ζώνη παραγωγής στην Ισπανία, υπάρχουν 18.000. Άρα η αντιπροσωπευτικότητα είναι 17,5% της Ισπανίας, ενώ 13,8% μόνο για τη Γαλλικία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επεξεργασίας και μεταποίησης, ε, τα στοιχεία, τα, τα, ο κύκλος εργασιών, στην Ένωση των 27 είναι με βάση στοιχεία της Eurostat, ο κύκλος εργασιών είναι 18 δις ευρώ. Η Ισπανία έχει το 1 τρίτο από αυτά. Το 1 τρίτο, 6 δισεκατομμύρια, ενώ το 25% του συνόλου της Ευρώπης των 27 το έχει η Γαλλικία. Μιλάμε λοιπόν για μια χώρα και μια περιφέρεια όπου η μεταποίηση έχει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, τα αλλιεύματα. Αν λάβουμε υπόψη τα τρία βασικά δεδομένα ε, αλίευση, υδατοκαλλιέργεια και επεξεργασία. Αθροιστικά βλέπουμε ότι πρώτο για τα αλίευματα σύμφωνα με τα στοιχεία της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ της Ένωσης για τους 27 της Ένωσης ανερχόμαστε στα 7 δις ευρώ, η υδατοκαλλιέργεια 3 δις ευρώ και η μεταποιητική βιομηχανία στην Ευρώπη των 27 18 εκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τώρα της κατάστασης στον μεταποιητικό κλάδο. Εγώ θα επικέντρωνα την ε, παρέμβασή μου στο ότι είναι επικεντρωμένη σε παράκτιες ζώνες που εξαρτώνται ιδιαίτερα από την αλία. Επιπλέον ότι η Ένωση θέτει στο εμπόριο πάνω από 12 εκατομμύρια τόνους προϊόντων αλίας και υδροκαλλιέργειας που κάνουν την Ένωση πρώτη αγορά στον κόσμο μπροστά από την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ. Επιπλέον, η Ένωση, στην Ένωση της Ένωσης υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνικής βιομηχανίας και τρίτων χωρών. Υπάρχει μια υψηλή εξάρτηση από τις, εξαγωγές, εισαγωγές. Πάνω από το 60% των προϊόντων που, που μπαίνουν στο εμπόριο στην Ένωση προέρχεται από εισαγωγή. Υπάρχει επιπλέον μια τάση μείωση των αλλιευμάτων, ενώ υπάρχει μια πίεση στα αλλιεύματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαχειριστικά μέτρα. Άρα πρέπει να αναζητηθεί μια προσπάθεια βιωσιμότητας των πόρων. Να σας πω επιπλέον ότι υπάρχει μια υψηλή ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας προϊόντων της θάλασσας, υπάρχουν γύρω στις 4.000 επιχειρήσεις στην Ένωση, επεκτείνεται η δατοκαλλιέργεια, εμφανίζονται νέα προϊόντα με την έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει μια επέκταση του προϊόντος σε παγκόσμιο, του, των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυξάνονται οι νέες συνήθειες ε, και οι απαιτήσει του καταναλωτού, ποιότητα, αλλαγή, ε, ε, ενημέρωση, ζητήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα ζούμε σε μια οικονομική και νομισματική αλλά και ενεργειακή περιοδικά κρίση. Ποιοι πρέπει λοιπόν να είναι οι στόχοι της ε, κοινή πολιτικής αλληλεία κατά την απόψή μας. Πρώτον, να εξασφαλίσει ότι υπάρχει υπεύθυνη αλληλεία, φθηνό και βιώσιμο εμπόριο, να ενισχύεται η υπεύθυνη συμμετοχή και η βιώσιμη συμμετοχή όλων των, ε, όλης της αλυσίδας στην αλλήλευση με περιβαλλοντικά και κοινωνικονομικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσει την κοινοοικονομική βιωσιμότητα και την μελλοντική αναγωνιστικότητα του κλάδου, της ελεία και της υδατοκαλλιέργεια, αλλά και των μεταποιητικών των προϊόντων μεταποίηση. Ποιε είναι οι προτάσει μα ε, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, η Επιτροπή έλεγε ότι ο, η αξία της παραγωγής της μεταποίησης ήταν 18 δις. Το διπλό δηλαδή του, συνόλου των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας και της αλίας. 3 και 7 δισεκατομμύρια αντίστοιχα. Κατά την άποψή μας, δεν μπορούμε, ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι η πράσινη βίβλα για τον μεταποιητικό τομέα ε, αγνοήθηκε. Διαβάστε το ίδιο το, την ίδια την πράσινη βίβλο και θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες παράγραφοι όπου ε, γίνεται μια μικρή μνήμα στην κοινοτική βιομηχανία μεταποίησης. Για να είναι επιτυχής η κοινή αλληλευτική πολιτική ωστόσο πρέπει να συνδέεται απόλυτα με το τι συμβαίνει στην αγορά από την άποψη του εμπορίου και των αγορών και να διαμορφώνεται ε, ε, ε λειτουργώντας με ενοποιημένη προσέγγιση του αλεκτικού κλάδου, ε, στον οποίο θα παρεμβαίνουν η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση και το εμπόριο. Και στον τελευταίο αυτή περίοδο και με εισαγωγέ όπως προέκυψε σαφώς από τις συζητήσεις. Αν λάβουμε υπόψη την κοινή πολιτική αλληλείας και, την κοινή οργάνωση, και τις κοινές οργανώσεις αγοράς μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μείωση των ε, αλλιευμάτων, μια ισχυρή εξάρτηση από τις αγωγές, μια εξέλιξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης, μια σημαντική επέκταση της υδατοκαλλιέργειας, αύξηση της κατανάλωσης, αλλαγή των ε, καταναλωτικών συνηθιών, και επέκταση του εμπορίου των προϊόντων αλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι παράκτιες χώρες θέλουν να παίξουν ρόλο στον τομέα αυτό. Σημαντικό ρόλο. Άρα, οι νέες προκλήσεις ε, πρέπει να εξελιχθούν νομοθετικά και κανονιστικά μέσω της κοινή οργάνωσης αγοράς, εξασφαλίζοντας δίκαια εισοδήματα, αλλά σταθεροποιώντας αυτόχρονα και τις αγορές. Άρα, για σήμερα πρέπει να εξασφαλίσουμε υπεύθυνη και βιώσιμη αλία και εμπόδιο και να εξασφαλίσουμε το μέλλον όλων των κρίκων της αλυσίδας και της μεταποίησης και εμποδία των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Αν μπούμε στην εμπορική πολιτική, εισαγωγέ, προμήθεια, πρόσβαση στην αγορά και καθεστώ ανταλλαγών με τρίτε χώρε, θέλω να σα πω ότι οι επιχειρήσει του μεταποιητικού κλάδου αλληλεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτε στις, ε, στα ανεβοκαταβάσματα τη προμήθεια. Άρα για να εξασφαλιστεί τακτική προμήθεια αλληλευτικών προϊόντων, οι επιχειρήσει τη Ένωσης πρέπει να προσφεύγουν σε εισαγωγέ. πρέπει να διαθέτουν ε, κατάλληλο προϊόν, επαρκέ προϊόν για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στην αγορά. Οι εισαγωγέ στην αγορά της Ένωσης εξαρτώνται από τις ε, ε, εκφορτώσεις στην Ένωση, που δεν είναι αρκετές όπως γνωρίζουμε. Επιπλέον πρέπει να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκή τροφοδοσία σε πρώτη ύλη που επιτρέπει στη μεταποιητική βιομηχανία να αυξήσει την παραγωγή και να δημιουργήσει θέσει εργασία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει για, όλους τους, για επιχειρήσεις, τόσο κοινοτικέ επιχειρήσει, όσο και επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Επίσης, η κατάσταση των πόρων στην Αλία πρέπει να αντιμετωπίζεται με μια συνεκτική πολιτική μεταξύ των πολιτικών συντήρησης ό,τι αφορά το μέγεθος και, της, και την αλίευση, αλλά ταυτόχρονα η Ένωση πρέπει να προωθεί και να παροτρύνει την υπεύθυνη και βιώσιμη αλία μέσω εμπορικών πολιτικών, που θα εξασφαλίζουν, όπως είπα, την βιωσιμότητα των ε, επιχειρήσεων μεταποίηση στην Ένωση. Γι' αυτό το λόγο παίζει σημαντικό ρόλο, παίζουν σημαντικό ρόλο οι εισαγωγές, ώστε να συμβάλλουν στο ευρύτερο πλαίσιο της αλληλευτικής πολιτικής της Ένωσης. Κατά την άποψή μας πρέπει να προσπαθήσουμε σε ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες πρόσβασης της αγοράς που αποτελεί σημαντικό για την, σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη αλία. Πρέπει να υπάρχουν απαιτήσει στήριξη των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού όλων των επιχειρήσεων του κλάδου κοινοτικών και τρίτων χωρών. Σε ό,τι αφορά την υγιεινή, την, ε, ε τις εργασιακές σχέσεις, τη φορολογική, την περιβαλλοντική και την ε, αλληλευτική Και πρέπει να πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η τήρηση τη νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, ιδίω αυτών που προέρχονται από τρίτε χώρε. Το λέω αυτό διότι η, συχνά η, όταν γίνονται συμφωνίες και εμείς που ταξιδεύουμε και βλέπουμε άλλες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι οι απαιτήσει Τις όλαφοι του FVO δεν ε, είναι οι ίδιες. Το ίδιο φορά και τις ε, περιβαλλοντικές. Από την 1η πρώτη του 10 η νομοθεσία για την παράνομη ελεία πρέπει να καλύπτει και τρίτες χώρες. Μιλώ για χώρες ε, της ΑΣΕΑ, που μετέχουν στο ΑΣΕΑΝ, χώρες του Ειρηνικού, όπως Παπουαζία, Νέα Γουινέα κλπ. Οι συνθήκε πρόσβαση της αγοράς, ε, τώρα σε ό,τι αφορά η έλεγχη που έκανε η FVO, η υπηρεσία, δηλαδή η κτηνατική υπηρεσία της ε, η Γενική Διευθυνσάμκο της πρέπει να γίνονται και σε επιχειρήσεις και σε εκφορτώσεις. Πρόκειται για επιθεωρήσεις ε, που θα γίνονται σε εγκεκριμένε ε, δομέ με εγκεκριμένε ομάδε. Πρέπει να εξασφαλίζονται ότι οι εισαγωγές και οι πρώτοι ύλοι που πηγαίνουν στην αγορά τηρούν τις, όλες τις απαραίτητες νομοθεσίες σε όλη τη διαδικασία μεταποίησης. Ισοδύναμα με αυτά που απαιτούνται για την κοινωνική παραγωγή. Εμεί κάναμε μια, μια μελέτη για την αγορά του τόνου πριν από δύο χρόνια, όπου το 65% των προϊόντων πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών και ε, για τον τόνο δεν τηρούσαν καμία από τις ε, κοινοτικές ε, προϋποθέσεις, στην επισήμανση, στην, ε, στην επεξεργασία κλπ. Εμείς θέλουμε τον ανταγωνισμό, ξέρουμε να ανταγωνιζόμαστε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε, αλλά πρέπει να τηρούν όλοι τους ίδιους κανόνες και να υπάρχει παρόμοια επαγνύπρινση, παρόμοιος έλεγχος παντού. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά πρέπει η πρόσβαση να είναι ισορροπημένη. Το καθεστώ εμπορικών ανταλλαγών με τρίτε χώρε, αν δεν πρέπει να, να, είναι υποφελέ για τρίτε χώρε ει βάρο τη κοινότική νομοθεσία, όπω ε, για τον τόνο. Αν γίνεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζει την αρχή τη κοινοτική προτίμηση. Αυτή η αρχή υπάρχει μόνο επί χάρτου. Εμεί ζητούμε σε όλες τις συμφωνίες που πραγματοποιούνται να δίνεται, να γίνεται ε, παρακολούθηση, να υπάρχει έλεγχος θέτοντας ως στόχο της συμφωνίας ακριβώς αυτή τη μελέτη. Ταυτόχρονα ζητούμε να γίνονται μελέτες αντικτύπου που θα είναι και σοβαρές και σωστές και δεν θα έχουν στόχο να στηρίζονται σε κάποιες πολιτικές ε, ψευδής, ψευδούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα προϊόντα ανεξάρτητα προέλευση να στηρούν την κοινοτική νομοθεσία. Όχι όπω έγινε πριν ένα χρόνο όταν μία περιοχή απειλάγει απόλυτα από την εφαρμογή των κανόνων προέλευση, ενώ ταυτόχρονα πήρε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά, στην Ευρωπαϊκή αγορά χωρίς καμία ε, ε, χωρίς κανένα αντισταθμιστικό μέτρο. Με μια μελέτη αντικτύπου που κανένα άποψή μου και για να τα πω με, ευγενικά, με ευγενικό τρόπο δεν είχε και πολύ ουσία ούτε ήταν και πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρή. Στα πλαίσια των εμπορικών ε, διαπραγματεύσεων ε, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ένωσης και των χωρών με τι χώρες ΑΚΕ, με χώρες του Ειρηνικού, Παππού, Αφίτζη, με το γύρο της Δόχα πρέπει να υπάρχει μια ε, ισχυρή υποστήριξη των αλληλευτικών προϊόντων της κοινοτικής Ένωσης. Τα συμφέροντα του κλάδου της μεταποίησης στρεβλώνονται σοβαρά αντίθετα από αυτά που έγραψε ο κύριος Μπαρόζο, ο οποίος σε μία επιστολή είπε για να είστε πιο αντιπροσωπευτικοί, για να είστε πιο ανταγωνιστικοί, να πάτε στην Παπούα και να αφήσετε τους 12.000 εργαζόμενούς σας στα κρύα του Λουτρού. Αν αυτή είναι η άποψη της Επιτροπής και του κυρίου Μπαρόσο, νομίζω ότι δεν ενισχύουμε την απασχόληση στην Ένωση. Αν μη τι άλλο, αυτό που ζητάμε είναι η κοινωνική πολιτική να έχει συνέπεια σε όλους τους κλάδους. Να υπάρχει μια κοινωνικο-οικονομική και ανταγωνιστική βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας στην κοινότητα. Για να τελειώσω τώρα θα σας έλεγα ότι κατά άποψή μας πρέπει να βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της, ε, του κλάδου μας που λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο σε, έναν διεθνοποιημένο, σε μια διεθνοποιημένη αγορά. Πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την κοινωνικονομική βιωσιμότητα του κλάδου σε ένα διεθνές πλαίσιο. Επίσης, το, σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι η κοινωτική βιομηχανία πρέπει να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που να είναι ε, ένα πλαίσιο που θα είναι συνεπές με τις υπόλοιπες κοινωτικές πολιτικές, θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δεν μπορούμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή να μας λένε πηγαίνει τα παράγεται στην Κεντρική Αμερική, για παράδειγμα, ή στην κοινότητα των άνδρων και μετά να ανοίγει μια άλλη αγορά, τη Ταϊλάνδης για παράδειγμα, που να καλύπτει το 30% της κοινωνικής αγοράς ε, στον τόνο χωρίς να υπάρχει καμία αντιστάθμιση. Εμείς ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε ότι εμφανίζονται προϊόντα από αγορές ε, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ε, Ταϊλάνδης κλπ. χωρίς καμία ε, πολιτική αντιστάθμιση. Συμπερασματικά. Η μελλοντική κοινωτική πολιτική, ε, κοινή πολιτική αλληλεία θα πρέπει να ενισχύει το εμπόριο, την βιώσιμη αλληλεία, να τηρεί το κανονισμό για την παρανομή αλληλεία. Δεν μπορεί να υπάρχουν 200, τόν, δολάρια τόνου διαφοράς ανάμεσα στην παραγωγή του νόμιμου τόνο από εμά από την, τον παράνομο τόνο των ε, πλοίων από την Ταϊβάν. Να ενισχύουμε την ανταγωνιστική του κλάδου και τη βιωσιμότητα τη μεταπαιδευτική μηχανία, να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα τη αγορά να εξασφαλίσουμε την προμήθεια σε πρώτη ύλη τη μεταποιητική κοινοτική βιομηχανία, να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα εξασφαλίσει την ισορροπία μακροπρόθεσμα όλη τη αλυσίδα στην αλληλευτική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα και η επιστημική ασφάλεια των προϊόντων, επαγρυπτώντα για την αχνηχνευσινόμενότητά και να ενισχύσουμε την ερευνητική δραστηριότητα του κλάδου. Ταυτόχρονα ζητάμε ήδη κανόνε ανταγωνισμού, να υπάρχουν ήδη κανόνε ανταγωνισμού για όλου του ε, εργαζόμενου, για όλε τι επιχειρήσει στον κλάδο, να ενισχυθεί σωστή κοινοτική προτίμηση και να υπάρξει μια ενεργή προάσπιση των ευρωπαϊκών αλληλευτικών προϊόντων. Η μεταρρύθμιση τη κοινή πολιτική ε, αλληλεία με τον τρόπο αυτό πρέπει να παρέχει μηχανισμού και μέσα που θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κοινοοικονομική βιωσιμότητα ε, του κλάδου και της μεταποίησης και που θα είχε συνέπεια, ως συνέπεια ένα καλύτερο μέλλον όλου του κλάδου της Ελίας. Έχω πολλά πράγματα να σας πω κύριε Πρόεδρε ακόμα, αλλά Ελπίζω κάτι τη διάρκεια των συζητήσεων να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ και... θέλει λόγο? Α, κύριε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Αλληλείας θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου αφενός τα εισοδήματα των αλληλείων να οργανωθούν με τρόπο αποτελεσματικό και φυσικά ότι η μεταπιτική βιομηχανία και οι σχετικοί απασχολούμενοι ε, θα έχουν δυνατότητα επιβίωσης, αλλά αφετέρου θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύεται και η φύση και τα ψάρια τα οποία όλοι χρειαζόμαστε να εξακολουθήσουν να υφίστανται αναφέρθηκε ότι το 88% ε, αφορά υπεραλίευση. Δεν ακούσαμε τίποτα σήμερα για την υπεραλίευση. Θα ήθελα να μας πείτε αν ε, και εσείς συμφωνείτε με τα αριθμητικά στοιχεία αυτά ή αν έχετε κάποια διαφορετικά στοιχεία. Είπατε ότι η νέα οδηγία για τον έλεγχο είναι αστείο. Θεωρείτε ότι κατά το παρελθόν ο έλεγχος δεν έγινε με τον δέοντο τρόπο, γιατί νομίζω ότι αν ήταν σωστός ο έλεγχος δεν θα είχαμε τόσο καταστροφικούς αριθμούς, ε, αριθμητικά στοιχεία σήμερα. Αναφέρθηκε ότι είναι πολύ χαμηλές και οι τιμές. Μπορεί, αλλά στην τελική ανάλυση η τιμή που φτάνει στον καταναλωτή είναι πάρα πολύ υψηλή. Άρα αναρωτιέμαι, τι δεν πάει καλά στην αλυσίδα και να εξηγήσω τι εννοώ. Τα τελευταία χρόνια στην Γεωργία αντιμετωπίσαμε παρόμοια προβλήματα σε ό,τι αφορά το γάλα. 18 σέντ ε, δίνονται στον παραγωγό, ενώ του χρειάζονται 38 για να επιβιώσει. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην αλληλεία. Να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό εκ νέου. Πού βρίσκονται τα δύναμα αυτά σημεία. Γιατί από τη μία έχουμε υπερεαλίευση, από την άλλη δεν μπορεί να επιβιώσουν οι αλείς και κατά τρίτον ο καταναλωτής υποχρεώνεται να καταβάλει τόσο, υψηλό, τόσο υψηλή τιμή για το ψάρι που τελικά δεν μπορεί να το φάει όσο θα έπρεπε κάθε εβδομάδα. Κάτι δεν πάει καλά όμως. Μίλησα προηγουμένως για το θέμα της υδατοκαλλιέργειας. Θα ήθελα να επαναλάβω όσα είπα. Αν θεωρήσουμε ότι οι εισαγωγές στρεβλώνουν την αγορά μας, γιατί λοιπόν δεν επικεντρωνόμαστε στην Ευρώπη πιο πολύ σε υδατοκαλλιεργίες, προκειμένου να έχουμε δικά μας ψάρια, τα οποία θα ακολουθούν τα δικά μας πρότυπα. Είπατε ότι είναι πολύ ψηλά τα κριτήρια για την δημιουργία τέτοιων μονάδων. Δεν υπάρχει όμως και κάποιο τέτοιο σχετικό περιφερειακό σχέδιο για το πώς θα προωθούνται οι ιδιωτοκαλλιέργειες. Ύστερα αναφέρθηκε ότι τα φιλέτα τηλάπια και παγκάσιου ε, πληρούν λίγο πολύ τα ίδια κριτήρια όπως και τα δικά μας προϊόντα. Και θυμάμαι μια φορά που είχα φάει κάτι τέτοιο Διάβασα ότι το Υπουργείο προειδοποιεί ότι ε, ενδεχόμενο ερυθρό χρώμα του φιλέτου της τηλάπια θα μπορούσε να υποδεικνύει η χρήση του παγορευμένου μονοξιδίου του άνθρωκα. Και σε παρόμοιες εξετάσεις προέκυψαν τέτοια στοιχεία και ε, το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα φιλέτα αυτά. Δεν ε, μπορώ να πω, έχω μείνει άφωνη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε ίσως εσείς. ε... Λοιπόν, ο κύριος Καντέκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με αυτά που μας είπε ο κύριος Κέλλερ. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει τον κύριο Κέλλερ είναι ότι ξέρουμε ακριβώς ε, που, τι θέλει να πει. Είναι σαφής, έτσι, πολύ σαφής. Ε, έχετε πραγματικά το, ε, ε, το πλεονέκτημα να χαρακτηρίσετε από απόλυτη ειλικρίνεια και σαφήνεια υπερασπίζεστε πάρα πολύ καλά του επαγγελματίε του κλάδου σας, τους μεταπητές και τους χονδρέμπορους, είναι σαφέ. Τώρα, το λεχθέντος, δεν με πείσατε, γιατί κυρίω ε, οι προβλέψεις οι αριθμητικέ για το 2015. Ε, είναι ιδιαίτερα τυχαίε, θα έλεγα και δεν πρέπει να τις πάρουμε τις μετρητή. Και με βάση την εμπειρία μου Πρέπει να σας πω ότι ε, η δημιουργία μοντέλων ε, με κάνει δύσπιστο. Παρά τον τόνο του λόγου σας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αντίθεση με τα ποιητές παραγωγή. Απλά και μόνο θέλουμε να έχουμε όλοι όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ελία και επιτρέποντας ταυτόχρονα μια αποδοτική αλλαγή και μεταποίηση. Θέλω να σας ρωτήσω εξής κύριε Κέλλερ λοιπόν. Πιστεύετε, με βάση αυτά που είπα, ότι αυτά τα οποία είπατε και οι προτάσεις σας θα επιτρέψουν να διασφαλίσουμε τη μεταποίηση και τη χονδρική πώληση και ταυτόχρονα την επιβίωση ε, του, της Ευρωπαϊκής Αλίας μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε και εμείς και αυτό το ερώτημα θέλω να θέσω και σε εσά. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Σούζα. Δεν ξέρω. Μπατίστα δε Σούζα. Ναι. Κύριε Σούζα. Μιλάτε για κοινοτική προτίμηση για τα μετεποιημένα προϊόντα. Ε, η ερώτησή μου είναι εξή. Κατά την άποψή σα, τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. αν ολοκληρωθεί ο κύκλο τη Δόχα με την υφιστάμενη βάση, πράγμα το οποίο είναι πιθανό να συμβεί και που προβλέπει ε, ε, ε, τους η τελωνική δεσμή τώρα από το 23% να πάνω στο μείον 6%. Και λαμβάνοντα υπόψη και κάποιε άλλε προτιμήσει, έτσι. Τι πιστεύετε, μάλλον το πω διαφορετικά, πιστεύετε το μοντέλο του καθεστώτος εισαγωγής Καθώ εισαγωγικών είναι θεμελιώδες πρόβλημα, είναι κοινό πρόβλημα για τους αλληλεί, για τους ηχθειοκαλλιεργητέ και για τους μεταπητέ. Αφορά κάποιου, ειδικά ή όλους. Γιατί αυτό το ερώτημα θα το θέσουμε και ίσω το μπορούσατε να μας απαντήσετε από τώρα. Αυτές τι παρατηρήσει θέλω να κάνω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σβαρέα έχει το λόγο. Μπαρέα. Νομίζω ότι το επίκεντρο ε, τον προβληματισμό μας είναι το κατά πόσον είναι απαραίτητες οι εισαγωγές. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία ακούσαμε από τη μεριά των μεταποιητών και από τη μεριά των... Ε, και μέσα καταναλωτές, οι εισαγωγές είναι απαραίτητες. Πρέπει όμως να δούμε πού μπαίνει η κοινωτική αγορά και το πώς. Πώς θα είναι ανταγωνιστική, ε, πώς θα βρούμε νέες, νέους τρόπους διάθεσης, πώς θα υπάρξει αυτορύθμιση της, της αγοράς, πώς θα ξατομικευθούν οι επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνοντα και τι μεταποιητικέ, με ε, τον καταναλωτή στο επίκεντρο, παρέχοντάς τους εγγύησεις, όπως είπε η κυρία Ρόντους Άρα και τιμές και προτιμήσεις. Και αυτό σε συνδυασμό μια εσωτερική αγορά που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ε, κοινωνικά χαρακτηριστικά, α, βιωσιμότητα ε, των αγορών, των αλλιέων, του περιβάλλοντος. Το να λέμε το κατά πόσον είναι αρνητικές θετικές εισαγωγές δεν βοηθά στον προβληματισμό οι εισαγωγέ φαίνεται ότι είναι απαραίτητε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το στοιχείο και επομένω να επανατοποθετήσουμε τον προβληματισμό μα, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τι δυσάρεστε συνέπειε, τι οποίε όλοι αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόβιν έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αριθμιστικά στοιχεία φυσικά τα οποία μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αναγκαζόμαστε να προβούμε σε τόσο υψηλές εισαγωγές για να καλύψουμε τις ανάγκες της συζήτηση, της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να μειωθούν οι εισαγωγές. Υπάρχουν και θέματα υπεραλίευσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εξαγάγουμε τα αποτελέσματα, τις συνέπειες της υπεραλίευσης στην Ένωση. Μία ερώτηση έχω να κάνω για την οικολογική και βιώσιμη αλληλεία, η οποία είναι ασφαλώς εξαιρετικά κρίσιμη για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Ωστόσο, από τις παρουσιάσεις του κυρίου Κέλλερ και των άλλων, ε, λείπει ένα στοιχείο. Μιλήσατε για το μέλλον, για το μέλλον της ζήτησης ε, των καταναλωτών. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία, ξέρετε, μένεται και στην ε, Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία, στη ΣΥΠΑ και στη Γερμανία, φαντάζομαι. τα ψάρια τα οποία εισάγονται από, την, από υδατοκαλλιέργειες ή από την ιστορική παραγωγή δεν θα πρέπει να κατανεμηθούν, να γίνει διάκριση, γιατί φυσικά η αλληλεία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και οικολογική. Αυτό είναι το οποίο ζητούν οι καταναλωτές σε τελική ανάλυση. Μία ερώτηση λοιπόν προς τον δόκτωρα Κέλλερ. κοιτώντας τα νομικά μέσα για την εισαγωγή αλευτικών προϊόντων, αν δεν εφαρμόζονταν, αν ήταν ανοιχτές και ελεύθερες οι αγορές, θα προτιμούσατε ένα τέτοιο καθεστώς, δηλαδή να επικρατούν ιδιωτικές ε, πρωτοβουλίες ιδιωτικών ε, οργανώσεων για την επισήμανση των βιώσιμων προϊόντων. Ποια είναι η θέση σας. Για αυτά τώρα που μας είπε ο εκπρόσωπος ε, από τη Σκοτία για το σκουμπρί, το οποίο εξάγεται Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά. για τη ρέγγα που εξάγεται. Είναι σημαντικό το θέμα αυτά. Και επίσης να δούμε τι ζητούν και οι καταναλωτές. Οι ενώσεις οι δικές σας θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου και το σκουμπρί και η Ρέγκα να καταστούν και πιο ελκυστικά προϊόντα για την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί το 60% των ε, αλληλευτικών ε, προϊόντων του σκουμπριού στην ε, Σουηδία χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Ο Σολομός καλλιεργείται και είναι ελκυστικό προϊόν. Τι λοιπόν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα των προϊόντων αυτών και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα είχαμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε και τις τιμές. Γιατί αφενός ε, η παραγωγή και η αλήθεια δεν παίρνουν τα χρήματα για, το, για τα τους, αλλά και οι καταναλωτές πληρώνουν υπερβολικά υψηλές τιμές. Άρα ίσως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει για να αυξηθεί η αξία του προϊόντος τελικά. Κλείνοντας. Μία ερώτηση ακόμα προς την μεταποιητική βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα τα παράνομα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που είναι γνωστό. Πώς ε, θα μπορούσε να αντιδράσει η μεταπητική βιομηχανία στο φαινόμενο αυτό σε ό,τι αφορά τα παράνομα αυτά αλλιεύματα. Τι μπορείτε να κάνετε για τη μεταποίησή τους. Ευχαριστώ κύριος Πρεσέδο. Ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, μιλητές. Ε, κύριε Κέλλε, νομίζω ότι θέσατε ε, ειλικρινά ε, τις απόψεις και για το ρόλο της ΕΕ των αγορών. Όμως μετά από αυτή τη χρηματοπιστωτική κρίση και την οικονομική κρίση που όλοι γνωρίσαμε, να εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα, οι αγορές είναι τέλειες, τι να σας πω, νομίζω θα έπρεπε να έχουμε λίγο περισσότερη ταπεινοφροσία. Ο μίλησε για τη σημασία αξιών όπως ε, η ασφάλεια, ε, τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε στο επίκεντρο των προβληματισμών μας για την αλία και να μην ε, περιμένουμε να δράσουν αυθόρμητα οι αγορές. Τώρα να σας πω κάτι και ε, όσον αφορά αυτά τα οποία ακούσαμε ε, και από τον κύριο Τεσούζα. Εγώ έρχομαι από την ίδια περιοχή και πρέπει να σας πω ότι ε, η, ε, η, η βιομηχανία κατασκευής κονσέρβας θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την συνολική πολιτική, αν θέλουμε μια λύα για την Ευρώπη. Επίσης πιστεύω ότι όταν μιλάμε για προάσπιση της βιομηχανίας, δεν, είμαστε, δεν ασκούμε προστατευτισμό, είναι παγκοσμιοποιημένη η βιομηχανία. Και αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφάλεια, σε υγεία, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την έρευνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνδυασμένα όλα αυτά με κοινωνικές πτυχές κτλ. Άρα, ε, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία τίθεται σε εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα ε, νόμιμο και θεμητό να πιστεύουμε ότι τα πρότυπα θα πρέπει να είναι τα ίδια ανεξάρτητα με το που κατασκευάζονται αυτά τα προϊόντα. Και μην ξεχνάμε ότι λαμβάνονται διάφορε απόφασει σε διεθνή φόρα για το θέμα αυτό. Και δεν μπορούμε εμεί να βρισκόμαστε στο περιθώριο ε, όλων αυτών των αποφάσεων στο μέλλον. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο ε, για λόγου χρόνου δεν αναφέρθηκε. Για λόγους χρόνου δεν αναφέρθηκε. Η σχέση βιομηχανία εμπορίου. Και αυτό αποτελεί μέρο προβληματική στον αλληλευτικό τομέα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διασπορά. Ε, στη βιομηχανία η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη. Αλλά σε εμπορικό επίπεδο τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι σχέσει ανάμεσα στο εμπόριο και στη βιομηχανία και θα θέλαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτά τα στοιχεία γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κ. Φεραίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκαλεσμένους μας, να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας και για την σαφήνεια την οποία επιδείξατε στις παρουσιάσεις αυτές. Γιατί οι σαφές και για μας ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η τοποθέτησή σας. Και αυτό με τη σειρά του καταδεικνύει ότι μιλάμε για έναν τομέα ο οποίος ε, διακρίνεται από την παράλληλη ύπαρξη ε, διαφορετικών συμφερόντων πολιτική αλληλείας, οι σχετικές εμπορικές πολιτικές και το πώς εφαρμόζονται, το πώς διαμορφώνονται, δεν είναι και αυτές ε, ουδέτερες, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την κατάρτιση και την κατάσταση των πολιτικών αυτών. Το πρόβλημα έχει ήδη αναφερθεί. Η πολιτική, η αλληλευτική και η σχετική εμπορική πολιτική κατά την εφαρμογή τους που ουσιαστικά μόνο μειονεκτήματα ε, συνεπάγονται για τον κλάδο. Οι τιμές για το τελικό προϊόν για τον καταναλωτή παραμένουν οι ίδιες, ίσως και να αυξάνονται και υπάρχει παράλληλα μια σειρά εγγυήσεων ε, για την υγεία οι οποίες δεν επαρκούν. Και έχουμε χάσει αυτά τα δύο άκρα, αν θέλετε, της αλυσίδας. Και στο εσωτερικό κάπου υπάρχει το κέρδος ε, στη μεταπητική βιομηχανία τους με μεγάλους εμπόρους οι οποίοι κερδίζουν από την πολιτική αυτή. Αναφέρεται ότι οι εισαγωγές δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς την εθνική παραγωγή, αλλά ότι υπονομεύουν σε πολλές περιπτώσεις τις ε, τιμές για την εθνική παραγωγή. Και τελικά αυτό επηρεάζει τα περιθώρια μεταξύ των κρίκων της αλυσίδας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας είναι σημαντικοί και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη γιατί όλοι παίζουν το ρόλο τους. Το θέμα είναι όμως να υπάρξει και μια πιο δίκαιη κατανομή των ε, υπεραξιών αυτών στο εσωτερικό της αλυσίδα μεταξύ των κρίκων. Αυτό ζητάμε και ο συνάδελφος ε, Καντέκ. Είπε και στις δύο συνεδριάσεις ότι δεν είναι δυνατόν η αλληλευτική πολιτική να θυσιαστεί στο βωμό του διεθνούς εμπορίου πολύ σωστά. Αλλά τι γίνεται στην πράξη. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στα λόγια και σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να αναγνωρίσει τι γίνεται και στα θέματα τα ελληνικά. Έχουμε και άλλα μέτρα για τη σκηνή, για τα ποτομισιακό καθεστώς. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, του παραγωγού σημαίνει ότι χρειάζονται κανόνες και για την, το εμπόριο και ότι η απορρίθμιση, όπως παρουσιάζεται ως τώρα, αν θέλετε αμφισβητεί όλα αυτά τα στοιχεία, την προστασία του καταναλωτή, του παραγωγού, των αποθεμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαραντίκα, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές για, την, για τις ομιλίες τους. Νομίζω ότι μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις όλοι έχουμε σχηματίσει μια πιο συνολική εικόνα των προβλημάτων αυτών. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι εμείς από τη σκοπιά της Ευρώπης και μάλιστα από τη σκοπιά της Επιτροπής μας ε, έχουμε ξεκαθαρίσει και συνοψίζω αυτή τη στιγμή ότι, ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το βασικό ερώτημα είναι αν θέλουμε μια ολοκληρωμένη ελευτική πολιτική ή όχι. Αν θέλουμε ένα, ε, μια ελεία στην Ευρώπη ή όχι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και στη συνέχεια ε, πιστεύω ότι δεν υπήρξε αντίφαση ανάμεσα στις ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα. Ο καθένας έχει συγκεκριμένη θέση σε ένα τομέα και αυτές οι θέσει είναι συμβατέ. Εγώ όμω θέλω να κάνω την ερώτηση. Δεδομένου ότι τουλάχιστον τα μέλη της Επιτροπής μας είμαστε υπέρ μια ολοκληρωμένης πολιτικής ε, αλληλευτική και για ένα, μια ευρωπαϊκή αλληλεία έτσι ώστε στο μέλλον τουλάχιστον να μην εξαρτώμεθα από τρίτε χώρε ανάμεσα στι άλλε ε, μα. Ήθελα λοιπόν να σα πω ότι σε επίπεδο ε, παραγωγής, ε, παραγωγών ε, ε, πραγματικά έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι δεν αντέδρασαν έγκαιρα ε, στις αλλαγές ε, της κατανάλωσης κτλ. Ότι πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να είναι αποδοτικοί και να έχουν μια βιώσιμη πολιτική αλλά και μια πολιτική σαφής σε επίπεδο μεταποίησης όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού, ε, χρειαζόμαστε εισαγωγέ, είναι σαφέ ότι στην αγορά απαιτούνται νέα προϊόντα. Υπάρχουν, υπάρχουν μελέτε ε, για τι συνήθειε των νέων κτλ. Ε, ε, ανάγκη σε φιλέτα κτλ. Συμφωνώντας λοιπόν ότι απαιτείται μια συνεκτική πολιτική στην Ευρώπη, σε επίπεδο όλων των αποφάσεων που λαμβάνουμε, ότι απαιτούνται πραγματικοί έλεγχοι Ω προ τα προϊόντα ε, τα εισαγόμενα, γιατί και αυτό είναι άλλη καταγγελία που ακούσαμε και ακούμε διαρκώς σε όλες τις επαφέ μας με τους διάφορου εκπροσώπου των επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν, αναγνωρίζοντα όλα αυτά, να σα ρωτήσω το εξή. Κανείς από εσά δεν αναφέρθηκε στο θέμα ποιότητα. ως παράγοντα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Αλίας. Πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν στα πλαίσια του καθορισμού μιας συνεκτικής και πιο διαφανούς πολιτικής στον τομέα της αλίας. Έτσι ώστε οι αποφάσει να μην λαμβάνονται μόνο ε, με βάση πολιτικά συμφέροντα, γιατί αυτό το διαπιστώνουμε και εμεί πολλέ φορέ στην Επιτροπή μα. Εσεί λοιπόν πιστεύετε ότι η ποιότητα, όπως ακριβώς έγινε και σε άλλους τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράγοντα ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ελίας. Τόσο επίπεδο παραγωγή τόσο και επίπεδο μεταποίηση. Δεν θα μπορούσε η ποιότητα να μας αυξήσει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έγινε σύγκριση με το κοτόπουλο, ναι. Μπορεί να θέλει τι τιμέ ο καταναλωτή, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το γάλα και με άλλα προϊόντα. Και όμω, η διάκριση του ευρωπαϊκού προϊόντος από τα υπόλοιπα προϊόντα γίνεται με βάση την ποιότητα. Ενώ να γνωρίζουμε ότι χρειάζονται και εισαγωγέ. Εσεί λοιπόν πώ βλέπετε, πιστεύετε στην ποιότητα ω παράγοντα ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο παγκοσμίων αγορών. Και κάτι άλλο. Τι, τι θέλετε από την Επιτροπή μας ε, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού τομέα που χαρακτηρίζεται από ευθύνη και έλαβε αποφάσεις και λαμβάνει αποφάσεις για τη διαχείριση. Πρόσφατα, στη χώρα των Βάσκων, μετά από πέντε χρόνια που δεν μπορούσαμε να ψαρέψουμε την, ε, το γάβρο, την αντσούγια και ε, ανεξάρτητη ποσοστώση διαχειρίζεται ε, το σχέδιο ίδιο το τομέα. Αποφασίζοντα το πότε, πόσο θα αλλιεύσει ε, και σε ποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ε, να γίνει και αυτό ο τομέα ανταγωνιστικό, διατηρώντα την ποιότητα, διατηρώντα τι τιμέ, διατηρώντα τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Θέλω λοιπόν να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανεί άλλο το λόγο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω κι εγώ ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε το βασικό θέμα. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στη μεταποίηση. Και νομίζω ότι κανεί δεν διαφωνεί με αυτή την παρατήρηση. Έγιναν διάφορε παρεμβάσει και από τον τομέα τη μεταποίηση και αυτό είναι λογικό βεβαίω. Ε, για παράδειγμα, ένα εκπρόσωπο τη Γερμανία ε, έχει την αλφα τοποθέτηση, γιατί ακριβώ στη Γερμανία γίνεται μεταποίηση και όχι η αλία. Ε, αλλιώ βλέπουν το θέμα οι χώρε παραγωγή και αλλιώ οι χώρε μεταποίηση. Εντάξει και ο κύριος Κέλλερ ε, τον ξέρουμε, έτσι, ξέρουμε το χαρακτήρα του, θέλει να μας προκαλεί. Οπότε δεν μας πειράζουν αυτά που λέει. Σαφώς υπάρχει ένα τμήμα του τομέα τη μεταποίησης που έχει διαφορετικά αιτήματα από τους αλληλείς. Και σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Το θέμα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρούμε ισορροπία και για τις εισαγωγέ. Γιατί, κοιτάξτε, ο κύριος Μαξουίν είπε κάτι με σαφήνεια. ε, όσον αφορά την εξάρτηση από τις αγωγές. Και δεδομένου του λόγου που ανέπτυξε, ε, δεν θα μας οδηγήσει κάτι τέτοιο σε χαμηλές τιμές ή σε ε, εφοδιασμό ε, της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Να μην σας αναπτύξω τους λόγους, το ανέπτυξαν οι ομιλητές καλύτερα από μένα. Πάντως, εγώ θέλω να κάνω μια σειρά από ερωτήσεις. Κύριε Βιέιτες. Μίλησε ε, για ε, κανονικό εφοδιασμό και ασφάλεια εφοδιασμού. Ρωτώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια εφοδιασμού όσον αφορά τις πρώτες Το σύστημα τελωνιακών ποσοστώσεων, δεσμολογικών ποσοστώσεων. Η διαδικασία που έχει καθοριστεί στα πλαίσια της κοινή οργάνωσης αγοράς δεν αρκεί. Τι λείπει ε, και γιατί. Δεύτερο θέμα στο οποίο θα θέλω να αφαιρθώ. σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Βιέδας και άλλοι εκπρόσωποι, σε σχέση με ε, τις πρώτες ύλες ε, και τα λοιπά και τους ελέγχους. Δηλαδή, για τη μεταποίηση της κονσέρβες ε, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα πρότυπα. Και αναφέρθηκε στο 65% κονσέρβας τόνου. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Και πώ λειτουργεί το σύστημα αυτό, κυρίω έναν των τρίτων χωρών, γιατί σα είπατε σαφώ ότι τόσο όσον αφορά τι εγκαταστάσει όσο και τα σκάφη δεν γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, ίσω και λόγω έλλειψη προσωπικού, αλλά είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι άμα θα φάμε το μπαγκάσιο θα, θα πεθάνουμε. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριο Βιέτε. Άρα λοιπόν, ποιο έχει την ευθύνη και πώ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Όσον αφορά του κανόνε καταγωγή. Πριν από λίγα χρόνια, ε, ξέρουμε τι έγινε. Ε, γιατί λοιπόν, τι, γιατί υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τους κανόνες προέλευσης ή καταγωγής ε, και τι θα γίνει τώρα με το θέμα αυτό, πώς θα συνεχίσουμε. De acuerdo con un tema que ha dicho el señor que me parece que es importante, sobre todo. Τώρα κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε, το οποίο είναι σημαντικό, που έχει να κάνει με την νομική ασφάλεια των επιχειρήσεων. Μερικέ φορέ ε, ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωτική πολιτική, ε, όπως για παράδειγμα με τη ΣΥΠΑ και με τι γενικευμένε προτιμήσει. ε, και με, τη, με την κατάσταση εταιριών ε, ε από την Ισπανία κυρίω κτλ. Ε, το, ε, το ανέφερε και ο κ. Μπαρόσο. Προβαίνουν σε κατάσταση και μετά ε, ξέρουμε τι έγινε με την εμπορική πολιτική ε, και με ορισμένες ασιατικές χώρες. Δηλαδή γίνεται μετακατάσταση και μετά δεν έχω καμιά εγγύηση για τότε θα εξακολουθήσουν να έχουν το ίδιο σύστημα. Και τώρα να δώσω το λόγο α, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στους ομιλητές. Και, και κοιτάξτε και οι ομιλητές του πρώτου πάνελ μπορούν να πάρουν το λόγο αν το επιθυμούν. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέιτς ε, της Γενικής Διεύθυνσης Μάρη και μετά θα πάρει το λόγο κύριε Γκαρθία. Έχετε το λόγο. Ε, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση σήμερα το πρωί και ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία σημειώσαμε και με προσοχή για τις αναλύσεις μας, για την ε, αναθεώρηση της ε, ΚΟΑ σε ό,τι αφορά την αλληλευτική πολιτική. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία. Αρκετοί ομιλητές μίλησαν για τη μεγαλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή. Θεωρούμε ότι η αναθεώρηση της ΚΟΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο πολύ εστίαση στον τομέα αυτό γιατί επί του παρόντος ε, εστιάσατε στις υποχρεωτικές πληροφορίες, στις ε, μεθόδους ε, παραγωγής των αλλιευμάτων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επεκταθούν οι πληροφορίες αυτές, να υπάρχει περιθώριο και για εθελοντικές, αν θέλετε, προαιρετικές πληροφορίες προς τους καταναλωτές βάσει ε, κάποιων βασικών αρχών. Ακούσαμε, για παράδειγμα, την ιδέα της οικολογικής επισήμανσης, η οποία αναπτύχθηκε σε ιδιωτικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά ιδιωτικά πρότυπα, ως επιτοπλίστων, ως σήμερα. Θέλαμε πέρσι να εισάγουμε τέτοια ε, κριτήρια για προαιρετικά στοιχεία τα οποία δεν πέρασαν όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μήπως θα μπορούσαν να ενσωματωθούν τα στοιχεία αυτά στα πρότυπα διάθεσης της αγοράς της ΚΟΑΣ, στην αγορά της, της ΚΟΑ. Επίσης εργαζόμαστε επισταμένα για το νέο αυτό παρατηρητήριο της αγοράς και το μέλλον, στο μέλλον ελπίζουμε να βελτιωθεί η οικονομική αντίληψη και για τους δύο τομείς, για τους οικονομικούς φορείς και για τους ε, φορείς παρατηρήσεις της αγοράς. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη η οποία θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για την υδατοκαλλιέργεια, και το κατά πόσον υπάρχει σχετική έμφαση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό το συζητήσαμε και χθες το απόγευμα, το συζητήσαμε ξεχωριστά και στην έκθεση του κυρίου Μιλάνα, άρα δεν θα το σχολιάσω και πάλι σήμερα. Έχουμε ένα τέταρτο μόνο. Περνάει ο χρόνο, δεν το κατάλαβα, πρέπει να φύγουν και οι διερμηνείς. Λυπούμε λοιπόν πολύ, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα, αλλά τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή. Θα ζητήσω λοιπόν από όλους όσοι θέλουν το λόγο τώρα να είναι σύντομοι. Κύριε Γκαρσία Φεραίρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις να σας πω για τη μελέτη αυτή της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, διότι αμφισβητήθηκε στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Δεν ξέρω αν παρανοήθηκα. Εγώ δεν είπα ότι οι τιμές δεν είναι χαμηλές, αλλά ότι άλλοι παράγοντες δεν λαμβάνονται υπόψη για το, τη μείωση των τιμών, ο κατακαιρματισμός του κλάδου, η στάση του καταναλωτή. Αν δείτε τη μελέτη ωστόσο, η μελέτη, και θα σας πω στα αγγλικά, η ανάλυση των κλάδων ε, δείχνει ότι εν γέννη δεν υπάρχει ζημία στον, στην κοινοτική παραγωγή από τις εισαγωγές όταν η εισαγωγή προκύπτει από την αδυναμία της κοινοτικής παραγωγής να καλύψει την ε, ζήτηση. Τώρα, για τους κανόνες ε, προέλευσης. Η Επιτροπή θεωρούσε ότι πρόκειται για νησιά που είναι απομονωμένα, εξαρτώνται από την αλληλεία, δεν έχουν επαρκή στόλο και ε, είναι καθαρά δραστηριότητα αναπτυξιακής βοήθειας. Σε άλλες αιτήσει η απάντησή μας ήταν αντική. Η Κομισιόν δεν έχει πρόθεση να έχει σε άλλη συμφωνία παρέκκληση των κανόνων προέλευσης, ιδίω εναντί χωρών της Ασίας. Μιλήσατε για την απομάκρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης σε τρίτες χώρες. Μιλώντας για ασιατικές χώρες. Ε, εμείς ξεκινήσαμε συζητήσεις με τη Σιγκαπούρη που δεν έχει όμως μεγάλη ε, σημασία. Καταλαβαίνουμε τη σημασία του κλάδου του, της ε, στην Ένωση. Όπως είπε ο κύριος Κέλλερ, τον ευχαριστούμε και αυτόν. Είναι διαστάσεις που λαμβάνουμε υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Να μιλήσω και στις για τις παρεμβάσεις της κυρίας Μπαρέα και της κυρίας Μπιλμπάου που μίλησαν για τις δυνατότητες αλλαγής συνθήκων για, το, τομέα της ποιότητας και της αλλαγής των, ε, της έμφασης της παραγωγής. Συμφωνούμε μαζί της. Με τις αλλαγές στον κανονισμό δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση ε, στην ποιότητα. Με την εξάλληψη των δασμών η ποιότητα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Μια τελευταία παρατήρηση. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά το άτομο. Δυόμιση. Κύριε Κέλλερ καταρχήν. Σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη αν σας προκάλεσα, αλλά μου ζητήσατε να μιλήσω με σαφήνεια. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω όμως, γιατί πολλές ερωτήσεις μου τέθησαν. Δεν ήταν η ΒΒΕΦ η οποία διαπίστωσε ποσοστό 88% υπεραλίευσης, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξέρετε ότι φυσικά πάντα αναφέρεται και η μέθοδος όταν αναφέρονται τέτοια αριθμητικά στοιχεία. Δηλαδή 88% όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο MSY, 30% όταν χρησιμοποιούμε την αρχή της πρόληψης. Αυτά τα αναφέρουμε για λόγους ειλικρίνειας. Αλλιώς τον έχει νόημα να κάνουμε τέτοιες ε, συγκρίσεις. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, συνεπή ε, και πιο αυστηρούς ε, ελέγχους. Αυτό που είπατε για την ε, κόκκινη τηλάπια αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς από την βιομηχανία, από τον κλάδο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί μετά από 8 χρόνια της εφαρμογής της οδηγίας για την επισήμανση έχουμε ακόμη ποσοστό 73% των προϊόντων που δεν ε, φέρουν τη σωστή επισήμανση. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει παρά μόνο με τον έλεγχο που είναι ελλειπής. Είπατε κύριε Καντέκ ότι δεν συμφωνείτε με τα αριθμητικά μου στοιχεία ε, και εντάξει το κατανοώ γιατί είναι δική μου η στατιστική αυτή, ο στατιστικός αυτός υπολογισμός. Αλλά να σας πω ότι θα σας προκαλέσει έκπληξη ότι δεν θα είναι 15 τα εκατομμύρια τόνοι αυτά που ανέφερα προηγουμένως σε πόσα χρόνια, θα είναι 18 εκατομμύρια και θα είναι πολύ πιο υψηλή η αριθμή αυτή. Θα το δείτε είπατε πώς μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των ε, αλλιέων και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν διοργανώνατε ένα σεμινάριο για την περαιτέρω διαμόρφωση της συνεργασίας αυτής. Επίσης, ακούσαμε μία ερώτηση για την επισήμανση. Φυσικά το MSC και το ISC θα αποτελέσουν τις ε, πιο επικρατούσες ε, σημάνσεις για το μέλλον και θα υπάρχουν και άλλες. Δεν θα υπάρχουν όμως καινούργιες ετικέτες, ούτε ευρωπαϊκές, γιατί δεν θα γίνουν αποδεκτές, θα έχουν επικρατήσει οι άλλες. Και κοιτάξτε τι γίνεται και με το αποτύπωμα σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, τα ύδατα. Θα δείτε ότι στην ευρωπαϊκή παραγωγή θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί μιλάμε για μικρές ποσότητες και αυτό το carbon footprint έχει να κάνει με μεγαλύτερες ποσότητες για την παράνομη αλληλεία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μας γιατί υπάρχει σχετική ρύθμιση, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον συνάδελφο Μαξουίν για τις πληροφορίες, την οδηγία για τις πληροφορίες για για τα τρόφιμα. Από το έτος 2012 θα πρέπει τα λιπαρά ψάρια να αναφέρουν στην ετικέτα τους το ποσοστό λίπους. Δηλαδή η ρέγατο, σκουμπρί, θα πρέπει να χρειάζονται κάθε τρίμηνο καινούρια επισήμανση γιατί αλλάζει αυτός ο ποσοστός λιπαρότητας αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν. Και ο καταναλωτής στην τελική ανάλυση θα πει «Ε, ας πάρουμε κοτόπουλο που ξέρουμε τι περιλαμβάνει τουλάχιστον σας». Παρακαλώ λοιπόν να τα λάβατε αυτά υπόψη και ε, σας προτείνω το, στο μέλλον να προτιμάτε το ψάρι. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά μας μένουν και εγώ θέλω και ένα λεπτό για να τελειώσω. Ο κύριος Μαξουίνη λοιπόν ε, θα μοιραστεί το χρόνο με τον κύριο Βίαιτε. Κύριε Μαξουίνη, σας παρακαλώ, ένα δευτερόλεπτο, πολύ λίγο. Σας δω συγγνώμη. Εν συντομία, αν και νομίζω ότι είπατε και εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των τομέων, γιατί και οι αλληλείς χρειάζονται τη μεταπληκτική βιομηχανία και αντίστροφα. Και ελπίζουμε και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η ευρωπαϊκή πολιτική να γνωρίσει ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους αλληλείς. Δεν μιλάμε για αλλαγή των σημάνσεων μία φορά το χρόνο, αλλά τέσσερις φορές το χρόνο για το ποσοστό λιπαρότητας. Ξέρετε, η ποιότητα του ψαριού αλλάζει με το μήνα. Δεν είναι τόσο σταθερό το προϊόν. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της μεταπητικής βιομηχανίας. Ρώτησε η συνάδελφος, έθεσε ένα θέμα για την ποιότητα. Είναι κρίσιμο το θέμα αυτό για την αλληλεία. Αλλά δυστυχώ το ερώτημα, στο, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αρνητική. Όχι. Οι αλληλείς δεν θεωρούν ότι ανταμείβονται για υψηλότερη ποιότητα προϊόντων. Και επικρατεί η άποψη ότι και με την οικονομική κρίση υπάρξε, υπήρξε μείωση της ποιότητας και ελπίζω αυτό να αλλάξει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σα ζητώ συγγνώμη να είσαστε πολύ σύντομοι. Σα παρακαλώ. Διαφορετικά θα τα πούμε σε διμερέ επίπεδο. Να προσπαθήσω να απαντήσω στα τρία ερωτήματα που ετέθησαν. Ε, πρώτα απ' όλα να σα πω ότι όσον αφορά το γύρο τη Δόχα, ε, ε, παγκοσμιοποίηση κτλ. Εδώ υπάρχουν ήδη ορισμένοι κανόνε, Ναι, είναι βασικό το πρόβλημα αυτό και αφορά ολόκληρο το τομέα του τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη αγορά στον κόσμο κονσέρβα τόνου και ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ισπανία με το 65%, ε, μετά ακολουθούν Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία και φτάνουμε στο 100%. Και επίσης η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε μέσω της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ ότι έχει αναθέσει μία μελέτη ε, που αφορά 40.000 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα έλεγα στην Επιτροπή ότι αν θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το κλάδο, αν θέλουμε να διατηρήσουμε, αν θέλουμε να χαρακτηριζόμαστε από ισορροπία και να μην καταστρέψουμε ε, την κοινωτική βιομηχανία και τι κοινωτικέ θέσει απασχόληση, ε, με την εξαίρεση ε, στου κανόνε, με την έλλειψη αυστηρότητα στου ελέγχου των προϊόντων τρίτων χωρών, όπου για παράδειγμα δεν γίνεται έλεγχος του προϊόντος που μεταποιεί το σκάφος ε, τρίτης χώρας, ε, και κατά πόσο βρίσκεται στου καταλόγου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υποχρεωτικό κτλ. Τώρα θα δούμε ε, με τι χώρε ΑΣΕΑΝ, κυρίω με την ε, Ταϊλάνδη, τι θα γίνει. Όσον αφορά ε, την παράνομη αλληλεία, ναι, ναι. εδώ πρέπει να δούμε τον ανταγωνισμό του τρίτου χωρών με τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να δούμε και τι επενδύσει κάνουν οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίε. Γιατί αποτελούν αντικείμενο ελέγχου απόλυτου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί. Αλλά δεν πάνε στην Νοτιοανατολική Ασία, στις τρίτες χώρες κτλ. Όσον αφορά ε, την ερώτηση του κ. Προσέντο, βεβαίω δεν θέλουμε προστατευτισμό. Αυτό που θέλουμε είναι ε, συμμόρφωση με του κανόνε, επαγρύπνηση και έλεγχο. Βιομηχανία και εμπόριο. Εδώ έχουμε δύο συνιστώσει και μία συνιστόσα είναι η διανομή. Από τη μια έχουμε πρώτη ύλη, ε, ποιότητα, ε, έτσι ώστε σε τελευταία ανάλυση να φτάνουν προϊόντα στον καταναλωτή, ώστε να είναι πιο ασφαλή και στην καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά ξέρουμε τώρα πώς δρούν τα μεγάλα καταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες διανομής. Ε, όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς, εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. Και βεβαίω και η εισαγωγή. και όσον αφορά την εκπρόσωπο, ε, το μέλος της Επιτροπής του Κοινοβουλίου από τη χώρα των Βάσκων, βεβαίως εμείς ε, ε, ταινίζουμε την Ευρώπη, κανόνες, πρότυπα κτλ. Αλλά όχι μόνο για ευρωπαίου Ευρωπαίους επιχειρηματίες και η ποιότητα βεβαίως και είναι σημαντική. Πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα, όλα αυτά έχουν ένα τίμημα. Άρα, μια πιο διαφανής πολιτική, είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, αυτό που χρειάζεται η μεταπητική βιομηχανία και σε περιόδους κρίσης πραγματικά Δυστυχώς βέβαια ε, η τιμή ε, έχει να κάνει με τα προϊόντα ποιότητας ε, και όχι με τις μεγάλες ποσότητες. Αυτό είναι γεγονός. Τελευταίο ζήτημα. Πρόεδρε, με ρωτήσατε για την ασφάλεια εφοδιασμού σε επίπεδο πρώτων Θα σας έλεγα ότι οι ποσοστώσεις αρκούν. Τώρα, στο μέλλον θα υπάρξει ανάγκη αύξηση Άρα δεν έχουμε ασφάλεια. Ε, πρέπει να ε, προβούμε σε εξορθολογισμό για να μπορέσουμε να, εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό σε προτεσίλες. Αλλά ελαμβάνοντα υπόψη την πορεία των αγορών, αυτό το οποίο απαιτείται είναι περισσότερο εφοδιασμό, περισσότερη προσφορά. Και ε, όσον αφορά τι τρίτε χώρε, ε, εδώ απευθυνόμαστε στις γενικές, στις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στις χώρες των κρατών μελών. Απαιτείται συντονισμό των ελέγχων στα σύνορα. Γιατί δεν γίνονται ε, σε ισότιμη βάση από όλου. Και οι κανόνες προέλευσης ε, ε βεβαίως εδώ ελπίζω η Γενική Διεύθυνση Trade, όπως είπε η κυρία Γκαρτία Φερέκ, να εξετάσει το ζήτημα. Ε, πρέπει να δούμε το θέμα της προβληματικής ε, στο συγκεκριμένο σημείο. Ε, και, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε αν πάνε οι πολυεθνικές στην Παππούα Γουινέα χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη και αυτό το αποδεικνύουμε και με την έκθεση που πραγματοποιήσαμε. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, που είχαν την καλοσύνη να με δώσουν λίγα λεπτά παραπάνω. Νομίζω ότι ε, η ακρόαση αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλους. Ε, συζητήσαμε ε, σε ευρία βάση διάφορα θέματα, τα οποία βεβαίως θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας για τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου και τους διερμηνείς, ε, τους εκπροσώπους του Γραμματείας, όλους. Ε, και πραγματικά να σας πω ότι Όσον αφορά του συντονιστέ, ε, μοιράσαμε τι αποφάσει που ελήφθησαν χθε στη συνεδρία των ιστών και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Επομένω, θεωρώ ότι ανακρίθησαν τα σημεία αυτά. Τελειώνω. Λίγη συνεδρία. Σα ευχαριστώ όλου για άλλη μια φορά. Ιδιαίτερα του διερμηνεί, λέει ε, η πρόεδρο, για τα λίγα λεπτά που μα έδωσαν. Θα τα πούμε την επόμενη συνεδρία. Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.